So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, Καλωσορίσατε στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε πιστεύω. Βλέπω χαρούμενα πρόσωπα μετά από μία εβδομάδα διακοπών. Αυτό σίγουρα καλό κάνει. Ελπίζω να επωφεληθήκατε. Το σημείο 1 είναι έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε δύο μικρές τροποποιήσεις. Καταρχήν οι ε, γνωμοδοτήσεις απαλλαγής της Utah Hawk. 8, 9, 10, 11, 12 και 13. Θα τις ψηφίσουμε πρώτα μαζί, on block, και μετά φτάνουμε στο σημείο 5 με τη δική μου γνωμοδότηση για το μέλλον των μεταφορών. Επίσης προτείνεται το 15 που είναι δική μου έκθεση. Μικρό θέμα. Είναι μια τυπική τροποποίηση. Να συζητηθεί ε, πριν το σημείο 14 που είναι της ε, κυρίας Κλάς. Ε, το δικό μου νομίζω θα το συστήσουμε γρήγορα διότι πρόκειται απλά για μια τυπική τροποποίηση. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Έχουμε όλες τις γλώσσες εκτός από στονικά, λετωνικά, μαλτέζικα, πορτογαλικά, σλοβένικα και σλοβάκικα. Αυτές οι γλώσσες δεν προβλέπονται. Το απόγευμα θα έχουμε Σλοβένικα όταν ο κύριος Πέτερλε μιλήσει για ε, το πρόγραμμα TREPS από τις 3 ε, μέχρι τις 4. Ε, από τις, 5 μέχρι τις 6. Επίσης θα εφαρμοστεί ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή τροπολογιών. Υπάρχει ένα σύστημα που ονομάζεται AT4AM, Authoring Tool for Amendments. Οι βοηθοί έχουν ενημερωθεί, υπήρχε και πρόσκληση για ε, μάθημα παρουσίασης, ε, η γραμματεία μπορεί να σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό, διότι 7 εκθέσεις ε, από αυτές που έχουμε στην ημερήσια διάταξη ε, θα ε, λειτουργήσουν με τον τρόπο αυτό. Δηλαδή μπορούν μόνο οι ηλεκτρονικά να υποβληθούν οι τροπολογίες. Έκθεση της κυρίας Παρβάνοβα για το Κοσλοντούι, η έκθεση της κυρίας Κλάσιατα για τα βιοκτώνα, του κυρίου Φιέλναρ για την ενημέρωση για τα φαρμακευτικά προϊόντα της κυρίας Εύανς, ε, του κυρίου Σλόβενς και της κυρίας Ματίας. Οι βοηθοί κυρίως λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουν να γίνει αυτό σύμφωνα, να υποβληθούν τροπολογίες σύμφωνα με το νέο σύστημα. Θα ήθελα να αναφέρω αυτό που όλοι διαβάσατε εκτελεστικός γραμματέας ε, της ε, Σύμβασης ε, του ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίματος. Για μένα αναπάντεχα ανακοίνωσε την την απόσυρσή του. Δεν θα ανανεωθεί η σύμβασή του που εκπνέει στις 30 Ιουλίου. Η Επιτροπή μας Θεωρεί θλιβερό το γεγονό αυτό, διότι είχαμε πολύ καλή συνεργασία μαζί του, ήταν πολύ ικανό. Ε, πουθενά δεν ε, λέει γιατί σταμάτησε, αλλά φαντάζομαι ότι η απογοήτευση για την Κοπενχάγη ε, τον άγγιξε βαθιά. Έχει δημιουργηθεί το νέο σώμα των ε, επιτρόπων μετά την έγκριση του ΣΕ στο Στρασβούργο. Υπάρχει μια σειρά ατόμων που θα ήθελα να αναφέρω, οι γενικοί ε, διευθυντέ του που μα είναι γνωστός. Θα γίνει Γενικός Διευθυντής για την ε, δράση κατά του κλίματος, ο κύριος και παραμένει Γενικός Διευθυντής της Γενική Διευθυνσή για το Περιβάλλον, ο Ρόμπερτ Ματλέν. παραμένει γενικός διευθυντής της ε, Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΓΟ και ο ε, Πέτερ Σέγγελ είναι γενικός διευθυντής ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια, που είναι επίσης τομέας που μας αφορά. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε επιστολή του Προέδρου της Κομισιόν Μπαρόσο προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων όσον αφορά την προστασία, την αλλαγή του κλίματος. Έχει οριστεί πρέσβης μας μια κυρία για το κλίμα στον υπόλοιπο, προς τον υπόλοιπο κόσμο ε, και το θέμα είναι βέβαια εάν θέλουμε να ε, εμείνουμε στις δεσμεύσεις μας ε, αναφέρεται δηλαδή ο στόχος του 30% ρητά στην επιστολή του κυρίου Μπαρόσο. Το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος μέσα Μαρτίου θα υιοθετήσει συμπεράσματα για τη βιοπικιλότητα και ε, ελπίζουμε να τεθούν στόχοι για τη διάσκεψη στην Αγκούη ε, φέτος τον Οκτώβριο, διότι η βιοπικιλότητα ε, θα είναι θέμα της χρονιάς 2010. Αυτές ήταν κάποιες ανακοινώσεις από τη δική μου πλευρά. Φτάνουμε στο σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών. Είχαμε τις συνεδριάσεις 13ης, 14ης, 15ης Ιανουαρίου και τις 25ης ε, έως 27ης Ιανουαρίου. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρηθεί ότι υιοθετήθηκαν. Και φτάνουμε έτσι στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης, ε, μια προφορική ερώτηση στην Επιτροπή μας. Έχουμε μία ερώτηση του συναδέλφου Μπάρτστας ε, για τα υλικά τα οποία έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Πρόκειται για ερώτηση προς την Επιτροπή. Ε, θα πρότεινα ο κύριος Στάς να μας παρουσιάσει το θέμα και ο Έρικ Πούτελε από τη Γενική Διεθνή ΣΑΝΚΟ της Επιτροπής θα απαντήσει κατόπιν. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα είμαι σύντομο. Έχει δυναμηθεί η ερώτηση, νομίζω είναι αρκετά λεπτομερής και θα ήθελα τώρα να ακούσω από τον εκπρόσωπο τη Εκκληστικής Επιτροπής ποιες είναι οι απαντήσει του. Ελπίζω να είναι καλέ απαντήσει και εξίσου λεπτομερείς. Στην ουσία περί τίνο πρόκειται. Υπάρχουν κάποια υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και στις περιπτώσεις αυτές χρειαζόμαστε διάφορες ε, νομοθετικές διατάξεις και αν δείτε και το website της Εκτελεστικής Επιτροπής υπάρχει ένα πολύ καλό ε, σκηνικό παρουσίασης της υπάρχουσας νομοθεσίας με ένα διάγραμμα που γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση όλων των υλικών και όπου αναφέρονται ακριβώς ποιοι είναι οι νόμοι οι οποίοι εφαρμόζονται στην κάθε περίπτωση. Το μεγάλο όμως πρόβλημα είναι ότι στην πράξη δεν υπάρχει μια έτσι ευρεία νομοθεσία, εκτός δηλαδή από τα πλαστικά και κεραμικά. Όμως άλλες ουσίες γύρω στις 10 δεν περιλαμβάνονται, δεν αναφέρονται. Και η νομοθεσία αυτή επαφείται πια για την εφαρμογή της στις χώρες μέλη. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα υλικά που με διάφορους τρόπους θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στο να ρωτήσουμε ή τόσο να θέσουμε κάποια ερωτηματικά σχετικά με την ασφάλεια για τα τρόφιμα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε ας πούμε, με περιπτώσεις όπως τα μελάνια. Τα μελάνια τα οποία εύκολα έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και θα μπορούσαν βεβαίως να δημιουργήσουν σοβαρές ε, σχολείες, σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν επίσης, υπάρχουν επίσης και κάποια προβλήματα σχέση με κάποια όρια, όρια που είχαν καθοριστεί παλαιότερα, χρονικά όρια. Πάντως νομίζω ότι εδώ χρειάζεται μια αναθεώρηση και θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Το θέμα αυτό είναι αρκετά σημαντικό που θέτω σήμερα, γιατί η, κατά κάποιο τρόπο έχουμε να κάνουμε μια εξέλιξη συνεχή, δηλαδή έχουμε τα διαφορά υλικά, έχουμε τα διάφορα μικροστοιχεία τα οποία και αυτά τέλο πάντων μπλέκονται εδώ, γι' αυτό ακριβώ το λόγο κατέθεσα αυτή την ερώτηση. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε στην ουσία με τέσσερι ερωτήσει. Αναμένω την απάντηση τη Εκκλαστική Επιτροπή, ώστε ενδεχομένω να σχολιάσω και εγώ το θέμα αυτό μαζί με του άλλου συναδέλφου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ε, συνάδελφε Στάση. Παρακαλώ η Επιτροπή να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να δώσω μια πλήρη απάντηση στον κύριο Στάς. Για το πρώτο ερώτημα να πω ότι η Γενική Διεύθυνση φέτος η DG Sanko θα ξεκινήσει την αναθεώρηση Τη ε, νομοθεσία που δεν έχει εναρμονιστεί πλήρω για αυτά τα θέματα. Θέλουμε να προβλέψουμε ένα σύστημα αποτελεσματικό για αυτή τη μη, εναρμονισμένη νομοθεσία. Ο κανονιστή προστατεύεται, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να αποφύγουμε και ένα περιττό φόρτο για τις αρχές και για τη βιομηχανία. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και την εξέλιξη τεχνολογίας σε αυτό το τομέα. Η εμπειρία μας δείχνει ότι με υψηλό αριθμό υλικών που έχουμε σήμερα, γύρω στις 10.000 που σε επαφή με τα τρόφιμα, χρειάζεται επαρκής χρόνος για να καθορίσουμε έτσι ένα κατάλογο διεξοδικό αυτών των υλικών. Θα μπορούσαμε λοιπόν να εξετάσουμε το ενδεχόμενο του positive listing μας με άλλε εναλλακτικέ λύσεις και θα προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη λύση ώστε να διασφαλίσουμε, όπως έλεγα, την προστασία των καταναλωτών και βεβαίως για να πετύχουμε και μια καλύτερη νομοθεσία που θα του προστατεύει. Αυτό ο νέο κανονισμό θα πρέπει να συνταχθεί μετά από μια αξιολόγηση επιπτώσεων σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο στους επόμενους 12 με 18 μήνες. Απαντώντας τώρα στην ερώτηση παριθμών 2, θα μπορούσα να πω ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι αυτά τα όρια είναι ένα κατάλληλο εργαλείο για την προστασία της υγείας του καταναλωτή. Αυτά τα όρια έχουν καθοριστεί μετά από επιστημονικές αξιολογήσεις κινδύνου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίμων και όσον αφορά αυτές τις ιδιότητες λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση κινδύνου όσον αφορά τη μετάβαση που έχει σημαντικές επιπτώσεις στον καταναλωτή. Όταν θα έχουμε λοιπόν νέες επιστημονικές ενδείξεις ή στοιχεία για την ποινότητα αυτών των ουσιών, τότε η υπηρεσία τροφίμων ε, θα ζητηθεί να επαναξιολογήσει. Προς το παρόν λοιπόν, οποιαδήποτε επιχείρηση που χρησιμοποιεί τον κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών και υλικών είναι υποχρεωμένη να κοινοποιεί την Κομισιόν αμέσως όταν είναι διαθέσιμα δηλαδή είναι επιστημονικά στοιχεία και να υποδεικνύει τον κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών. Απαντώντας τώρα στην ερώτηση 3 θα μπορούσα να πω ότι η εφαρμογή της άδεια για, για τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται και που, μάλλον, που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα έχει να κάνει με την προτινόμενη χρήση των υλικών αυτών. Η άδεια λοιπόν που θα πρέπει να δίδεται θα πρέπει να αφορά τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται και την αντίδραση που έρχονται αυτά τα υλικά όταν έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίμων θα κάνει και πάλι μια αξιολόγηση των κινδύνων και εάν υπάρξουν σημαντικά στοιχεία στην διαδικασία αδειοδότηση, τότε θα επιβάλλουμε κάποιου περιορισμού όσον αφορά την αδειοδότηση αυτών των ουσιών. Ενδεχομένω θα, θα είναι ε, περιορισμοί που θα αφορούν ε, το είδος τροφίμων με το οποίο θα μπορούν να έρχονται σε επαφή αυτά τα υλικά. Παρ' όλα αυτά, η διάδραση των υλικών αυτών με τη συσκευασία και τα τρόφιμα δεν μπορεί να είναι πλήρης, γιατί πολύ συχνά ο, ο παραγωγός των ειδών ε, συσκευασίας χρησιμοποιεί διαφορετικά είδη συσκευασίας και αυτό είναι μια γενική αρχή τέλο πάντων που υπάρχει στον ε, νόμο για τα τρόφιμα. Και απαντώντας τώρα στην ερώτηση 4, όλα τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα απαιτείται από τον νόμο να παρασκευάζονται σύμφωνα με μια χρηστή πρακτική ώστε να είναι βέβαιος ο παραγωγός ότι είναι ασφαλή τα προϊόντα του είτε μέσω εναρμόνισης βεβαίω ε, κοινωτικής νομοθεσίας, είτε όταν καλύπτονται πάνω από εθνική νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγός θα πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια των προϊόντων του μέσω της επιλογής των καταλήλων υλικών, μέσω ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής ώστε να μην παράγονται βλαβερές ε, ουσίες και υλικά μέσω ελέγχου του τελικού προϊόντος και αυτή η αρχή είναι εφαρμόσιμη για όλη την αλθίδα παραγωγής της συσκευασίας τροφίμων όλα τα υλικά, που, μάλλον όλα τα βήματα που λαμβάνονται θα πρέπει να είναι αντικείμενα τεκμηρίωσης από τον παραγωγό, θα πρέπει να ελέγχονται από τις εθνικές αρχές και τοξικολογικά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σχετικά με τα υλικά τα οποία μεταβιβάζονται, μεταφέρονται στα τρόφιμα και τα οποία δεν έχουν ακόμα εγκριθεί ή δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς την επικίνδυνοτητά τους. Γι' αυτό ακριβώς φέτος θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία αναθεώρησης σχετικά με την νομοθεσία που αφορά τα υλικά που έχουν σε επαφή τα τρόφιμα και δεν έχει εναρμονιστεί, τιμή εναρμονισμένη δηλαδή, και να περιλάβουμε κάποια υλικά όπως το αλουμίνιο, επιστρώσεις, υλικά που αφορούν επιστρώσεις και στην αναθεώρηση αυτή θα εξετάσουμε το κατά πόσο είναι απαραίτητο να περιλάβουμε περαιτέρω απαιτήσει λεπτομερείς όσον αφορά τα τοξικολογικά στοιχεία τα οποία θα είναι διαθέσιμα τέλο πάντων στην ε, διαδικασία παραγωγής ώστε να υπάρχει μια χρηστή πρακτική. Αυτή λοιπόν τη δικασία θα την ξεκινήσουμε και θα προσπαθήσουμε να δούμε επίσης και τη σχέση μεταξύ του REACH, αυτό το πρόγραμμα που όπως γνωρίζετε ε, εμπλέκει την Γενική Επιτροπή Περιβάλλοντος, επιχειρήσεων κτλ. και που αφορά όλες αυτές τις ε, ουσίες ώστε να υπάρχει μια διάδραση και με το πρόγραμμα REACH. Αυτά Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Υπάρχουν συμπληρωματικές ερωτήσεις, ε, κύριε Στάς. Ε, ε, ναι, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με την τελευταία απάντηση που έδωσε ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν, σε σχέση δηλαδή με την ερώτηση 4. Υπόθηκε επανειλημμένω κατά πόσο οι παραγωγοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάποιε έτσι χρηστέ διαδικασίε παραγωγή, αν θα πρέπει να είναι σχολαστική και τυπική στην εφαρμογή των ε, κανόνων κτλ. Όμως θα ήθελα να πω και επιμένω από αυτού ότι δεν θα έπρεπε, είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτό η παραγωγή. Και νομίζω ότι και οι δοξικολογικές δοκιμές βλέπω ότι για αυτές τις δοκιμές η Κομισιόν είναι κάπως διστακτική. Δηλαδή έχουμε 17 είδη προϊόντων. Προς το παρόν 15 ρυθμίζονται και ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με τα πλαστικά νομίζω ότι η νομοθεσία είναι επαρκής και υπάρχει ένα έγγραφο της αρχής του έτους από την Εκκληστική Επιτροπή όπου η Επιτροπή προβλέπει να λάβει υπόψη της τις υπάρχουσες οδηγίες και να τις ενοποιήσει υπό, μια, υπό ένα ενιαίο δηλαδή κανονισμό με ένα κείμενο διεξοδικό και πλήρες. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι θαυμάσια πράξη αυτή της Κομισιόν. Όμως, αυτός ο κανονισμός, εντάξει, για τα πλαστικά θα υπάρχει. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε αρκετά ναι αρκετές ελλείψεις. Επί παραδείγματι, χρωστικές ουσίες, διαλυτικά που χρησιμοποιούνται στη δικασία παραγωγή. τέτοια υλικά. Γι' αυτά λοιπόν τα υλικά η, η Κομισιόν στην πρώτη μου ερώτηση απαντά ότι θα υπάρξει μια νέα πρόταση κανονισμού τους επόμενους 12 με 18 μήνες. Ναι, αλλά έτσι το θέμα θα κρατάει χρόνια και το Κοινοβούλιο έχει υποβάλει, είχε υποβάλει το έτοιμο αυτό εδώ και πολύ καιρό. Θα έπρεπε λοιπόν να επιταχύνουμε κάπως τις διαδικασίες και Τέλος, θα μπορούσε να μας πει κάτι η Κομισιόν σε σχέση με τα μελάνια εκτύπωσης. Γιατί φοβάμαι ότι για τη δημόσια υγεία έχουμε πολλούς κινδύνους που έχουν αναδεχθεί πρόσφατα μάλιστα και από δημοσιογραφικές έρευνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ η συνάδελφος Κλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούω τώρα πώς ε, είναι χωρισμένες οι αρμοδιότητες ε, και με πιάνει φρίκι. Θα συζητήσουμε αργότερα την ε, οδηγία για τα βιοκτώνα. Μιλάμε εδώ για το μελάνι εκτύπωσης που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα. Και ρωτώ την Κομισιόν, μπορούμε να τα χωρίσουμε αυτά. Πώς θα αποφύγουμε επικαλύψεις στους διάφορους τομείς και πρέπει να αφαιρέσουμε κάτι από τα βιοκτώνα ε, διότι αργότερα θα ε, συμπεριληφθεί αυτό σε μια οδηγία σχετικά με τα υλικά τα οποία έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Πώς θα γίνει η διάκριση των ε, υλικών αυτών. Ευχαριστώ κύριε Σπούτελε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν μια απάντηση στον κύριο Στάση. Η μελλοντική νομοθεσία που προτιθέμεθα να υποβάλουμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο θα καλύπτει όλες τις ουσίες. Ξέρετε ότι πριν να προτείνουμε ένα σχέδιο κανονισμού στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο θα πρέπει να κάνουμε ένα impact assessment, δηλαδή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε όλες τις πιθανές ε, εναλλακτικές λύσεις, ώστε να δούμε το κόστος και το όφελος για τις επιχειρήσεις, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή είναι μια εργασία η οποία είναι μακροχρόνια, ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα που καλύπτει δεκάδες χιλιάδες ουσιών, με ένα σκέλος που εκπροσωπείται από την καινοτομία και ο κύριος Στάς μίλησε προηγουμένως για μικροστοιχεία και βρισκόμαστε ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα σε ένα τομέα πολύ καινοτόμο όπου η τεχνική και η επιστήμη συνήθως ε, συνεργάζονται και δημιουργούν συνεχώς νέες ουσίες. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε ώστε αυτές οι νέε ουσίες, αυτά τα νέα υλικά δεν θα έπρεπε να είναι επικίνδυνα για τους καταναλωτές και δυστυχώ δεν έχουμε ακόμα επαρκή επιστημονικά στοιχεία για αυτές τις νέες ουσίες. Εξάλλου, οι χώρε μέλη θα πρέπει να ελέγχουν την εφαρμογή των κανονισμών αφενός των κοινοτικών κανονισμών η οποία είναι πλαίσιο το γενικό δηλαδή κανονισμό όσον αφορά τελικά που έρχονται σε επαφή με το τρόφιμα και επίση και του επιμέρου κανονισμού όσον αφορά τι ομάδε ουσιών και ιδιαίτερα τι αναρμονισμένες. Αλλά επίση και τι ουσίε, οι οποίε δεν είναι αναρμονισμένες. Δηλαδή οι χώρε μέλη θα πρέπει να ελέγχουν όλη την εφαρμογή των ενδιαφερομένων αυτή τη χρηστή πρακτική των εργαστηρίων. Αυτό είναι ο ρόλος τους, αυτό θα πρέπει να κάνουν οι χώρε μέλη και θα πρέπει να μα κρατούν ενήμερους σε περίπτωση όπου υπάρχουν έλεγχοι και οι οποίοι καταδεικνύουν κάποια κενά ή ελλείψεις. Και αν ανακύψουν τέτοια κενά ελλείψει, θα πρέπει να πάρουμε και τα απαραίτητα μέτρα. Είναι αλήθεια ότι για τα μιλάνια κτύπωσης δεν έχουμε κοινοτική νομοθεσία, έχουμε όμω τι γενικέ γενικές αρχές του General Food Law που προβλέπει ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν να διαθέσουν ε, στην αγορά τρόφιμα τα οποία έχουν έρθει βεβαίω σε επαφή με τη συσκευασία μελανιών και είχαμε το 2007 κάποιο, κάποια υπόθεση στην Ιταλία όπου τα μελάνια διαπερνούσαν την συσκευασία τετραπάκ κάποιων τροφίμων, οπότε κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Και απαντώντας στην κυρία Κλάς να πω ότι έχουμε δύο είδη Τα βιοκτώνα καλύπτουν ένα σημαντικό, ένα συγκεκριμένο αριθμό προϊόντων μάλλον, που χρησιμοποιείται στην καθαριότητα και στην απολύμανση χεριών, υλικού που χρησιμοποιείται στην ε, βιομηχανία τροφίμων, στην κτηνοτροφία. Είναι ουσίες συγκεκριμένε που δεν καλύπτονται από την νομοθεσία που αφορά τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, που είναι μια νομοθεσία η οποία αφορά περισσότερο τα τρόφιμα στο σύνολό τους. Βεβαίως υπάρχει μια σχέση η οποία δεν είναι πολύ στενή αλλά παρόλα θα υπάρχει σχέση μεταξύ των ε, βιοκτώνων και των υλικών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και αυτή η σχέση, αυτός ο σύνδεσμος ήδη έχει ε, εισαχθεί στη νέα νομοθεσία για τα βιοκτώνα. Οπότε, αυτό καλύπτει δύο ιδιουσιών, όμως με ένα συντονισμό σε επίπεδο άδεια. Εκεί που υπάρχει επικάλυψη είναι ότι υπάρχουν υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα που χάρη στην κοινοτομία μπορούν να μετατραπούν σε βιοκτώνα. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε μια συσκευασία η οποία τέλο πάντων περιορίζει την ανάπτυξη βακτηριδίων όσο αφορά τα τρόφιμα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχουμε σχέση ε, ανάμεσα, μάλλον μεταξύ της νομοθεσίας βιοκτώνων και της νομοθεσίας που αφορά τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Οπότε θα μπορούσαμε να καθισχάσουμε την κυρία Στάση αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά είχα να πω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση πολύ σύντομα, Καρλ Σλούτερ. Αναφέρατε ότι είναι υποχρέωση των ε, κρατών μελών ε, να κάνουν τις δοκιμές και να εφαρμόσουν την νομοθεσία. Είπατε επίσης ότι θα σας δώσουν πληροφορίες. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πόσες δοκιμές έχουν κάνει τα κράτη-μέλη στις εκθέσεις που σας έχουν στείλει και πόσα προβλήματα βρήκαν. Τι ψάχνουνε στις δοκιμές αυτές. Είμαστε βέβαιοι ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται σωστά. Δυστυχώ δεν μπορώ να απαντήσω ε, για, στον αφορά τον αριθμό των τεστ που κάνουν τα κράτη-μέλη. Αλλά κάνουν τεστ. Ε, σε διαβεβαιώνω σε διάφορα επίπεδα στην αγορά, δηλαδή από τα εστιατόρια, από τα σούπερ μάρκετ, από τα σημεία πώληση παίρνουν τρόφιμα τα οποία έχουν συσκευαστεί όπως το νερό εδώ για παράδειγμα και βλέπουν κατά πόσο υπάρχουν ε, προβλήματα ε, μικροβίων. Ε, λοιπόν, γίνονται έλεγχοι στην αγορά, γίνονται έλεγχοι και στην εισαγωγή. Όταν εισαγωγείς εισάγουν πιάτα, κεραμικά, τηγάνια, κατσαρόλες, όταν εισάγουν πλαστικά, πυρούνια, ποτήρια, πιάτα, γίνονται έλεγχοι στην εισαγωγή. Και όταν οι έλεγχοι αυτοί δείξουν ότι δεν συμμορφώνονται τα προϊόντα αυτά στην κοινωνική νομοθεσία, τα προϊόντα αυτά στέλνονται πίσω στη χώρα προέλευσής τους. Σα διαβεβαιώνω λοιπόν ότι διεξάγονται έλεγχοι και στα σύνορα και στα κράτη-μέλη στην αγορά δηλαδή και στα εργοστάσια που παράγουν αυτά τα προϊόντα και βεβαίως όταν υπάρχουν μείζωνα προβλήματα σε προϊόντα τα οποία ήδη βρίσκονται στην αγορά ε, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες επισήμανσης στα πλαίσια ε, του δικτύου ταχείας επισήμανσης ε, για να ενημερωθούν τα διάφορα κράτη-μέλη που θα λάβουν αυτά τα προϊόντα για να αποσυρθούν τα προϊόντα από την αγορά. Συνεπώς ενεργοποιούνται πολλοί μηχανισμοί ώστε να αποσυρθούν από την αγορά αυτά τα προϊόντα όταν δεν ανταποκρίνονται στην νομοθεσία. Επίσης, οι επιθεωρητές μας της κοινότητας ε, ε, του, της υπηρεσίας των τροφίμων και της κινητικής υπηρεσίας πιστοποιούν κατά πόσο τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ε, την νομοθεσία για αυτά τα προϊόντα. Επισκέπτονται τα κράτη-μέλη για να δουν πόσοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί και πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία. Και αν ε, δεν επαρκεί. Αυτό αναφέρεται στις εκθέσεις και οι εκθέσεις είναι στη διάθεση του κοινού, είναι δημόσιες, μπορείτε να τις διαβάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το δύσκολο και πολύπλοκο αυτό ζήτημα για σήμερα και περνάμε σε μια μακρά σειρά ψηφοφοριών. Ελπίζω να έχετε όλη την ηλεκτρονική σας ε, κάρτα, διότι τις ε, τελικές ε, ψηφοφορίες θα τις κάνουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ λοιπόν να έχετε έτοιμες τις κάρτες σας. Είπαμε ότι τα 8 έως 13 θα τα ψηφίσουμε πρώτα. Πρόκειται για τις ε, απαλλαγές για τον προϋπολογισμό του 2008 ε, που προετοίμασε η συνάδελφος Γιούτα Χάοκ. Απαλλαγή 2008, Γενικός Προϋπολογισμός, ε, τμήμα Ρωμαϊκό 3. Τρεις ε, τροπολογίες υπάρχουν. Ε, παράγραφος 6, τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 της Γιούτα Χάουκ. Ε, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οριστική ε, ψηφοφορία για το θέμα αυτό, ε, ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας. λήξη της ψηφοφορίας. Είναι σαφές το αποτέλεσμα, 38 υπέρ, μία αποχή. Συγχαρητήρια στην Ιούτα Χάουκ για την έκθεση αυτή. Φτάνουμε στην, στις ψηφοφορίες για τις διάφορες υπηρεσίες. Ε, για τα χημικά. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν υπάρχουν ε, τροπολογίες. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την ε, έκθεση αυτή, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 41 υπέρ. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Περνάμε στην ε, ψηφοφορία για το ΕΚΠΕΝ. Μία τροπολογία της Utah Hawk. Ε, ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας που έχει και προφορική τροπολογία να διαγραφεί το ίντερνετ. Ποιο, ε, ε Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σύνολο της έκθεσης, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 40 ψήφοι υπέρ, μία αποχή. Περνάμε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Δεν υπάρχουν ε, τροπολογίες ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 41 ψήφοι υπέρ, μία αποχή, μία ψήφος κατά. Εγκρίνεται. Επόμενη ψηφοφορία αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ΕΜΕΑ. Δύο τροπολογίες Ψηφίζουμε την πρώτη της Γιούτα Χάουκ. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία του κυρίου Ούλμερ είναι όμοια με αυτήν της κυρίας Γιούτα Χάουκ. Δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σύνολο της έκθεσης. αρχή τη ψηφοφορία. Λήξη τη ψηφοφορία. 42 ψήφοι υπέρ, μία αποχή. Εγκρίνεται. Τελευταία ψηφοφορία αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Δεν υπάρχουν ε, τροπολογίες. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν για το σύνολο τη έκθεση, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη τη ψηφοφορία. 42 ψήφοι υπέρ, μία αποχή εγκρίνεται επίση Συγχαρητήρια στην Ιούτα Χάουκ για τις εκθέσεις της για την απαλλαγή ε, για το έτος 2008 της Κομισιόν και των διαφορών υπηρεσιών. Φτάνουμε στο σημείο 5. Φόρο μέλλον για τις μεταφορές. Πρόκειται για γνωμοδότηση. 39 τροπολογίες. Φτάνουμε στην τροπολογία 1, χωριστή ψηφοφορία έχουμε εδώ. Το πρώτο μέρος ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος. Ποιος είναι υπέρ του δεύτερου μέρους. Κατά αποχές ε, αποχές. Ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Ναι, σωστά το είδα. 18 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Εντάξει, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Α, απορρίπτεται. 21 ψήφοι υπέρ, 21 ψήφοι κατά. Ε, πολύ ε, μικρή διαφορά, καλά το είδατε, ε, μηδενική διαφορά. Τροπολογία 4 λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Α, όχι, εντάξει, αφέστε το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8-2β, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε, εντάξει. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Α, σαφές το αποτέλεσμα. 24 υπέρ, 16 κατά, μία αποχή. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 το πρώτο μέρος, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 21 το πρώτο μέρος, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21, το δεύτερο μέρος, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. 21, το δεύτερο μέρος, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται, ναι, είναι σαφές. 19 υπέρ, 25 κατά. Τροπολογία 18, το δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22, υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 18 κατά, με 4 αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5, ε, τροπολογία 17 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. κατά, αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Να ελέγξουμε την 27, εντάξει. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Α, εγκρίνεται. Συγγνώμη, εγκρίνεται. 27. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω εγκρίνεται, αλλά να το, να το επιβεβαιώσουμε. Ε, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 το πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο μέρος, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονικό έλεγχο για την 39 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Α, ναι, καλά το είδα. 24 υπέρ, 19 κατά, μία αποχή. Ε, ψηφοφορία για το σύνολο της έκθεσης ηλεκτρονική. Λήξη της ψηφοφορίας. 43 υπέρ, μία αποχή. Αυτή είναι λοιπόν η γνωμοδότησή μας προς την ε, Επιτροπή Μεταφορών για το θέμα εφόρο μέλλον για τις μεταφορές. Φτάνουμε τώρα στο επόμενο θέμα, το υπαριθμό 6, την ε, έκθεση της κυρίας Λιωτάρ για την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 Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Καταπίπτει. Όχι. Παρακαλώ. To ask the Commission to do research sur Το 11 ζητάει στην Επιτροπή να κάνει επιτόπου έρευνα στις χώρες παραγωγούς αυτοπληρώνων και να πει τι πώς μπορεί να βλάψει αυτή η παραγωγή την υγεία των Ευρωπαίων και ούτε η τροπολογία 11 ούτε 13 το κάνουν. Δηλαδή αυτή η τροπολογία ζητάει να γίνει έρευνα ακριβώς στο σημείο που υπάρχει η παραγωγή και συνεπώς η Επιτροπή θα έπρεπε να κάνει μια ανάλυση της, ε, της πιθανής βλάβης που μπορεί να προκαλέσει αυτό στη δημόσια υγεία. Εντάξει, να ψηφίσουμε λοιπόν την τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Ναι, άξιζε τον κόπο. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας η 15. Beendet. Ja, 23. 23 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. 16 ε, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι έχουμε την ίδια πλειοψηφία. Να το ελέγξουμε. 16, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Α, ακόμα πιο μικρή διαφορά. 22 υπέρ, 20 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. 17. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι είναι η ίδια πλειοψηφία, άρα εγκρίνεται. 18 υπέρ. κατά να ελέγξουμε τη 18 αρχή της ψηφοφορίας λήξη της ψηφοφορίας Ανάποδα. 20 υπέρ, 23 κατά. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 42 υπέρ, κανένας κατά. Συγχαρητήρια στην κυρία Λίοταρ για την έκθεσή της για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ιδατοκαλλιέργειας. Έχουμε μία ακόμα ψηφοφορία που αφορά το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Γεωσκόπησης του Βιτόριο Πρόντι. Ψηφίζουμε τις ε, τροπολογίες του εισηγητή. Ε, τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4, υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 26 κατά, απορρίπτεται. Φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία για την έκθεση αυτή, για το σύνολο της έκθεσης, ηλεκτρονικά, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 42 ψήφισαν, κανένας, 42 υπέρ, κανένας κατά. Ε, συγχαρητήρια στον Πιτόριο Πρόντι. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Γεωσκόπησης είναι πολύ σημαντικό. Η πρότασή μας ήταν ε, λοιπόν να ψηφίσουμε το σημείο 15 Πρόκειται για ένα τυπικό θέμα, δεν πρόκειται για τροποποίηση επί της ουσίας. Έχει να κάνει με την ποιότητα της νομοθεσίας. Το θέμα είναι ότι η Επιτροπή αλλάζει τη νομική βάση από απόφαση του Συμβουλίου σε οδηγία. Πρόκειται λοιπόν για νομοθετική διαδικασία με συμμετοχή του Κοινοβουλίου το 2004 στα πλαίσια του πακέτου υγιεινής η αρμοδιότητα της Κομμοσιών καθώς και το δικαίωμά της να αλλάζει κείμενα του Συμβουλίου επιβεβαιώθηκε από το Κοινοβούλιο. Η οδηγία του 2004 ε, από τον Ιούνιο του 2010 αντικαθιστά την παλιά απόφαση του Συμβουλίου και για να μην υπάρχουν νομικές ασάφειες θα πρέπει ε, να καταργηθεί η παλιά ε, νομοθεσία και να επιβεβαιωθεί η καινούρια. Το έγγραφο αυτό έχει να κάνει με τα έντυπα που όλοι οι εισαγωγείς ε, ζωικών ε, προϊόντων ε, θα πρέπει να χρησιμοποιούν. Η έκθεση κάνει ακριβώς αυτό. Καταργεί την ισχύ της παλιάς απόφασης του Συμβουλίου και επιβεβαιώνει την ισχύ της οδηγίας του 2004 από τον Ιούνιο του 2010. Πρόκειται λοιπόν για ένα τυπικό θέμα. Εγώ ως Πρόεδρος λοιπόν πρότεινα να ψηφίσουμε την έκθεση εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση. Και μήπως μπορούμε να ακούσουμε πολύ σύντομα την Κομισιόν και τους εσκιώδεις εισηγητές. Η Κομισιόν πολύ σύντομα όμως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι εσείς είπατε ό,τι χρειάζεται. Έχουμε να κάνουμε μια νομοθετική δράση για τη βελτίωση Τη διαφάνειας και της αφήνειας της κοινοτική νομοθεσία. Οι κανόνες εισαγωγή δεν αλλάζουν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Λαντομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Επιβεβαιώσατε αυτά που, είπα, που είπατε, ο, Σνάιντερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτό που αποφασίζουμε τώρα γίνει, ε, έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Πράγματι ήρθε η ώρα να ε, φροντίσουμε να υπάρχει νομική ασφάλεια, νομική βεβαιότητα, ασφάλεια δικαίου και θα πρέπει να καταργηθεί η παλιά διάταξη ώστε οι εισαγωγείς να ξέρουν τι ε, πρέπει να κάνουν. Ευχαριστώ πολύ, μπορούμε να ψηφίσουμε. Ωραία, δεν έχουμε άλλους να ζητούν το λόγο. Ψηφίσουμε λοιπόν ε, την έκθεση. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. ομόφωνα από ό,τι βλέπω, αποχές δεν υπάρχουν. Ε, ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε το σχέδιο νομοθετικού κανονισμού, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Χρειαζόμαστε το αποτέλεσμα, είναι σαφές το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν έχουμε ε, μια σαφή κατάσταση όσον αφορά το θέμα αυτό. Φτάσαμε λοιπόν στο θέμα 14 που είναι τα βιοκτώνα. Έχουμε εδώ έκθεση της κυρίας Κλάς και θα τη δώσω αμέσως στο λόγο. για να μας παρουσιάσει την έκθεση αυτή και κατόπιν θα τη συζητήσουμε. Παρακαλώ κυρία Κλάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε τα βιοκτώνα στην ημερήσια διάταξη και η ερώτηση του, Στάς, του κυρίου Στάς και η δική μου τελευταία ερώτηση έδειξε πόσο δύσκολο είναι το θέμα των ε, βιοκτώνων. Υπάρχουν πάντα επικαλύψεις και πάντα τίθεται το θέμα των ορισμών. Αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, ε, μπορείτε να είστε σίγουροι για ένα πράγμα. Ε, τα βιοκτώνα υπάρχουν σε πολλά προϊόντα, προϊόντα ε, καθαρισμού, προϊόντα συντήρησης ξύλου, ε, ε, προϊόντα καταπολέμησης, προϊόντα μειοκτώνα, παρασιτοκτώνα κλπ. Κάθε μέρα λοιπόν ερχόμαστε σε επαφή με τα βιοκτώνα. Στην έκθεσή μου το θέμα είναι η αναθεώρηση ε, της ε, οδηγίας για τα βιοκτώνα του 1998 και η μετατροπή της ε, σε κανονισμό. Συμφωνούμε για ένα πράγμα. Η υπάρχουσα οδηγία δεν αποδείχθηκε αποτελεσματική. Το πρόγραμμα αναθεώρησης έπρεπε το ε, πρόγραμμα ελέγχου έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, αλλά από ό,τι φαίνεται θα, θα κρατήσει μέχρι το 2015. Ο νέος κανονισμός ε, θα αναφέρεται στην ε, καταχώρηση και αδειοδότηση για όλα τα βιοκτώνα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προϊόντα με χαμηλή επικινδυνότητα θα εγκρίνονται από την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ΕΧΟ και οι υπόλοιπε ουσίε από τα κράτη-μέλη. Το, πρόγραμμα, το έγγραφο της Κομισιόν ε, θα πρέπει να ε, μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα και να απλοποιήσει την κατάσταση ώστε να είναι και πιο φτηνή η όλη διαδικασία, ώστε να μπορούμε να έχουμε σωστή προστασία από τα βιοκτώνα. Στη δική μου έκθεση έχω τονίσει τα σημεία. Καταρχήν, ε, τις ε, πτυχές ε, περιπαλλοντική προστασίας, κατά την αδειοδότηση, διάθεση στην αγορά και χρήση των διοκτώνων θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή της προφύλαξης. Και επίσης θα... Δεν θα πρέπει να λείπει η σύνδεση με, την Ευρωπαϊκή, με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Ήδατα. Η Κομισιόν προτείνει Ε, να αποκλείονται ε, τα προϊόντα με κάποια συγκεκριμένα ε, κριτήρια τις ουσίες που είναι επικίνδυνες για το ενδοκρινικό σύστημα 1α, 1β κλπ. Εγώ προτείνω και κάποια πρόσθετα κριτήρια ώστε να εφαρμόζουμε την αρχή της προφύλαξης και να λάβουμε υπόψη μας και τις περιβαλλοντικές πτυχές. Γι' αυτό αναφέρομαι στα PBT, τα VB και VP και τα ΠΟΠ. Ο ορισμός ε, των ε, των ουσιών για, ε, που προκαλούν ζημιά στο ενδοκρινικό σύστημα. έχω βασίσει τον ορισμό αυτών σε προηγούμενα νομοθετήματα, αλλά θα ήθελα να καλέσω την Κομισιόν μέχρι το 2015 να εκπονήσετε σχετικά κριτήρια και έχουμε επίσης τα CMR ε, κριτήρια της κατηγορίας 1β ε, καθώς ε, και την τοξικότητα ως κριτήρια για τις ουσίες αυτές. Η... Τα κριτήρια κατά τα άλλα αντιστοιχούν σε αυτά της, του κανονισμού για, τις, για τα φυτοφάρμακα και θα πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλα κριτήρια τα οποία χρειαζόμαστε, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης σε περίπτωση που η έκθεση ανθρώπων ή του περιβάλλοντος ε, απέναντι σε ε, δραστικές ουσίες ε, για παράδειγμα, η χρήση μιας ουσίας σε δόλωμα, αυτό θα πρέπει να αποτελέσει εξαίρεση. Θέλουμε να αποφύγουμε τους κινδύνους ε, για τους ανθρώπους ε, και για το περιβάλλον και ε, δεν θέλουμε να μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις οι οποίες να, δημιουργηθούν, να, να δημιουργούν κίνδυνο προς τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε με τις ευρείες εξαιρέσεις που θεσπίζουμε εδώ πέρα να μην υπονομεύσουμε το επίπεδο προστασίας. και για τις κατηγορίες 4, 14 και έως 19 ε, είναι πολύ σημαντική η δυνατότητα ε, άρσης της εξαίρεσης. Επίσης, ε, Έχουμε τα ανανοηλικά τα οποία χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά και αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στο σημείο 2 αναφέρομαι στην ε, προστασία των καταναλωτών. Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα προϊόντα που αγοράζουν ε, πληρούν ε, ενιαία κριτήρια ελάχιστον, μέγιστον ορίων. Τα πρότυπα ασφαλείας αυτά σημαίνουν ότι τα προϊόντα και των ε, Ευρωπαίων παραγωγών και ε, τα εισαγόμενα θα πρέπει να ε, πληρούν τα ίδια κριτήρια. Γι' αυτό προτείνουμε ένα σύστημα με αριθμό αδειοδότησης για όλα τα προϊόντα τα οποία έχουν τύχη μεταχείρισης από βιοκτώνα με εσωτερική και εξωτερική δράση, για παράδειγμα ε, έχουμε για παράδειγμα τα ε, συντηρητικά στις μπογιές, ε, έχουμε και, τα, και άλλα χημικά όπως είναι οι, τα, οι κουνουπιέρες και τέτοια. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιστοποιητικό ασφαλείας και οι καταναλωτές των βιοκτώνων θα πρέπει να ενημερώνονται για μη χημικές εναλλακτικές λύσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να ε, ενημερώνουν ε, τους καταναλωτές, θα πρέπει να γνωρίζει κανείς δηλαδή τι κάνει όταν χρησιμοποιεί βιοκτώνα, ιδιαίτερα όταν το κάνει στα πλαίσια της δουλειάς του. Σημείο 3 έχει να κάνει με την γραφειοκρατία. Η Κομισιόν προτείνει τα βιοκτώνα με χαμηλή επικινδυνότητα να εγκρίνονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ΕΧΑ. Ε, η CHA. Οι άλλε ε, θα πρέπει να εγκρίνονται από τα κράτη-μέλη με αμοιβή αναγνώριση. Αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, ποιο αποφασίζει αν ένα βιοκτόνο με χαμηλή επικινδυνότητα αν ένα βιοκτόνο έχει χαμηλή επικινδυνότητα ή υψηλή, η διάκριση αυτή δεν ορίζεται σαφώς και γι' αυτό εγώ προτείνω τη δυνατότητα ευρωπαϊκής αδειοδότησης για όλα τα προϊόντα. Γνωρίζω πολύ καλά ότι εδώ ζητάμε πολλά από την, ε, την ECHA, αλλά Η ECHA είχε μεγάλο φόρτο εργασίας με τον κανονισμό REACH Και γι' αυτό θεωρήθηκε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκή έγκριση για όλα τα προϊόντα. Αλλά κατά τη γνώμη μου το να ε, είναι αυτή η υπεύθυνη για όλε τι αδειοδοτήσει θα έχουμε ε, ευρωπαϊκή αγορά για τα βιοκτώνα. Όσον αφορά τις πληροφορίες για τα προϊόντα και τα ε, εμπορικά μυστικά, θα πρέπει να υπάρχει καλή ε, προστασία των δεδομένων και νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει πολύ καλύτερα κεντρικά. Και θα πρέπει να ισχύει το ίδιο χρονοδιάγραμμα με τον κανονισμό REACH. Όσον αφορά την αδειοδότηση, οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ε, για παράδειγμα τη συμπληρωματική αδειοδότηση για προϊόντα όπου έχει γίνει ε, μια μικρή τροποποίηση, όπως για παράδειγμα όταν έχει τροποποιηθεί το όνομα της ε, εταιρείας ή του προϊόντος. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιείται απλοποιημένη διαδικασία. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μειώσουμε το κόστος για τις επιχειρήσεις ε, κατά την αδειοδότηση των προϊόντων, ε, διότι τα βιοκτώνα χρησιμοποιούνται σε μικρές ε, ποσότητες. Όταν λοιπόν κανείς διαθέτει μικρές ποσότητες στην αγορά, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην επιβάλλουμε υπερβολικό κόστος στις επιχειρήσεις. Και δεν θα πρέπει το υψηλό κόστος για την για την καταχώρηση των προϊόντων να αποτρέπει τις επιχειρήσεις ώστε να ε, μην έχουμε ε, τόσο πολλά προϊόντα στην αγορά. Θέλουμε δηλαδή να προωθήσουμε την ε, ποικιλότητα όσον αφορά τα προϊόντα που διατίθονται. Ε, συνάδελφοι, το θέμα αυτό αφορά όλους μας. και εγώ έμαθα ότι σήμερα ότι στο, στην εκλογική μου περιφέρεια έχει ξεσπάσει ένα ιός σε νοσοκομείο όπου χρειάζεται, για την καταπολέμηση του οποίου χρειάζονται βιοκτώνα. Γι' αυτό είναι σημαντικό. να έχουμε ουσίες, βιοκτώνες, ε, για να μπορούμε να καταπολεμήσουμε ε, τα μικρόβια αυτά, τους ιούς αυτούς, τους οργανισμούς αυτούς που προκαλούν ε, επικίνδυνες αρρώστιες. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, τα βιοκτώνα για να έχουμε αποτελεσματικές απολυματικές ουσίες. Πρέπει όμως ε, να είναι αντικείμενο σωστής επαγγελματικής χρήσης οι ουσίες αυτές. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την εκπαίδευση των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις ουσίες αυτές, διότι αν δεν γίνεται σωστή επαγγελματική χρήση υπάρχει κίνδυνος της δημιουργίας ε, ανθεκτικότητας ε, στα μικρόβια. Τα βιοκτώνα είναι απαραίτητα, το γνωρίζουμε αυτό και ξέρω ότι και πολλοί συνάδελφοι από τις νότιες χώρες ασχολούνται με το θέμα αυτό λόγω το θέμα των παραστοχτών, των εντομοκτώνων. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των ε, βιοκτώνων, να μειώσουμε τους, τους κινδύνους και ελπίζω ότι θα έχουμε ε, καλές συνεισφορές από τις συναδέρφους ώστε να μπορέσουμε να εμείνουμε στο στόχο μας και να καταλήξουμε σε έναν καλό κανονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, εισαγωγή σου στο ενδιαφέρον αυτό θέμα. Πράγματι, από τη μία μεριά ε, έχουμε την ε, προστασία του περιβάλλοντος και από την άλλη την προστασία της υγείας. Και υπάρχει και το θέμα ότι υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις στον τομέα αυτών. Τα εξηγείς αυτά στην γνωμοδότησή σου. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, ο Ντάν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Γενικά νομίζω ότι η έκθεση αυτή θα κάνει την ε, νομοθετική αυτή πρόταση καλύτερη. Έχω κάποιες επικρίσεις, έχω και κάποιες θετικές παρατηρήσεις. Προτού φτάσω σε αυτές όμως ε, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τη διαδικασία, διότι μάλλον δεν φταίει ο εισηγητής, αλλά λάβαμε το δεν φταίει αλλά ε, λάβαμε πολύ αργά το κείμενο. Μας το είχαν υποσχεθεί πριν τα Χριστούγεννα, πολλέ αναβολέ έγιναν και ακόμα και σήμερα δεν έχω το οριστικό κείμενο στα δανέζικα. Έχω το κείμενο, αλλά έμαθα χθε ότι υπάρχουν κάποιε τροπολογίε οι οποίε υπάρχουν μόνο στα γερμανικά και το μεγαλύτερο μέρο του κειμένου το λάβαμε ούτω ή άλλω την Παρασκευή ή χθε ήταν. Εν πάση είχαμε πολύ λίγο χρόνο να εξετάσουμε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο θέμα. Είναι τεχνικέ οι τροπολογίε. Βέβαια, αυτό είναι πολύ καλό. Σημαίνει όμω ότι και εμεί θα πρέπει θα χρειαστούμε χρόνο να αξιολογήσουμε το κείμενο. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ε, ε, μεταφέρουμε την ε, προθεσμία για τις τροπολογίες. Μία εβδομάδα δεν αργεί, δεν έχω λάβει καν την οριστική μετάφραση των τροπολογιών. Πρόκειται λοιπόν για, μικρότερο, για λιγότερο από μία εβδομάδα για να εξετάσουμε αναλυτικά το κείμενο αυτό. Δεν ξέρω αν η εισηγήτρια ή ο πρόεδρος θα πρέπει να λάβει σχετική απόφαση, αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι απολύτως απαραίτητο. Ως προς το περιεχόμενο, καταρχήν να πω ότι Βρίσκω πολύ καλό ότι τονίζεται ότι πρόκειται για θέμα που αφορά το περιβάλλον και την υγεία ε, σε εξίσου μεγάλο βαθμό που αφορά την ε, ανταγωνιστικότητα, για παράδειγμα. Επίσης, ε, βρίσκω ότι είναι πολύ καλό ότι τονίζεται την αρχή της προφύλαξης. Αυτό σίγουρα ενισχύει την νομοθεσία. Γιατί όμως δεν μπορείτε να κάνετε το βήμα διότι στέλνετε τα σωστά μηνύματα ότι, ότι το θέμα αυτό αφορά την, ε, το περιβάλλον και την υγεία, αλλά αυτό δεν φαίνεται τελικά στο νομοθετικό κείμενο. Γιατί λοιπόν αντί απλά να στείλετε ένα μήνυμα δεν φροντίζετε να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα στο περιβάλλον και στην υγεία και αυτό ε, θα το πετύχουμε εάν έχουμε όχι ενιαία νομική βάση, να έχουμε μοιρασμένη νομική βάση, shared legal base. Ε, είμαι βέβαιος ότι θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες ε, για να έχουμε τριπλή νομική βάση ώστε να είναι θέμα που να αφορά και το περιβάλλον και την υγεία, ώστε να μην αφορά μόνο την ε, εσωτερική αγορά, να μην είναι νομική βάση, δηλαδή μόνο το άρθρο 95. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε διότι και το περιβάλλον και η υγεία είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και θέλουμε να λαμβάνετε υπόψη και κατά την εφαρμογή ε, της νομοθεσίας. Ελπίζω να είσαστε θετικοί απέναντι στην ε, δυνατότητα αυτή. Επίσης, όσον αφορά το στόχο, θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει περισσότερο να τονίσουμε ότι θα πρέπει να προστατεύονται ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες. Αυτό πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ήδη στο άρθρο 1. Άλλο σημαντικό που θέλω να τονίσω είναι ο ορισμός ε, των ε, ουσιών χαμηλής επικινδυνότητας. Ε, νομίζω θα συμφωνήσετε ότι είναι πολύ ασαφής ο ορισμός αυτός. Θα μπορούσαμε να τον κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Πάντως με τον υπάρχοντα ορισμό είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη η κατάσταση και είναι πολύ δύσκολο να κρίνει κανείς τι θα σημάνει αυτό στην πράξη. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη για πολύ πιο σαφή ορισμό, καθώς και η αντικειμενικότητα. Χρειάζεται λοιπόν εδώ... Χρειάζονται εδώ επιστημονικά στοιχεία, κυρίως από την Κομισιόν. Όσον αφορά τα κριτήρια cut-off, νομίζω ότι είναι πολύ καλό το ότι προτείνεται μια σειρά τροπολογιών που θα ευθυγραμμίσει την ομοθεσία αυτή με ε, την ομοθεσία που ισχύει για την προστασία των υδάτων. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να βοηθήσω να ε, σφίξω ακόμα πιο πολύ το κείμενο, πάντως είναι πολύ καλό αυτό. Όμως υπάρχει ένας τομέας όπου διαφωνώ λίγο με την γραμμή σας και έχει να κάνει με την εισαγωγή εξαιρέσεων, αποκλήσεων, τα derogations. Υπάρχει δυνατότητα απόκλησης ε, στο άρθρο 45. Δεν ε, θεωρώ ότι είναι απαραίτητες οι τρεις, ε, οι παρεκκλήσεις που εισάγετε εσείς, κυρία εισηγήτρια. διότι εισάγουμε έτσι τη δυνατότητα εξαίρεσης για τους παραγωγούς σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. βλέπω, δεν, φαίνεστε στενοχωρημένοι, αλλά θα πρέπει να το συστήσουμε αυτό περισσότερο εις βάθος. Ούτε θεωρώ ότι ε, συνάδει με την αρχή της προφύλαξης ε, το να έχουμε τόσες ε, εξαιρέσεις. Επίσης θέλω να αναφερθώ στη σχέση ανάμεσα στην έγκριση σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ECHA. Πρέπει να ομολογήσω ότι θα πρέπει να μελετήσω περισσότερο το θέμα για να μπορέσω να καταλάβω ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά είναι σαφές ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει ακόμα περισσότερο να γνωρίζουμε τι δυνατότητες βέτο, τι δυνατότητες ανησυχίες έχουν τα επιμέρους κρατημέλη. Αυτό το συζητήσαμε εις βάθος ε, και όταν συζητήσαμε την ε, νομοθεσία για την προστασία των υδάτων. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής. Θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια θέματα εις βάθος σε περίπτωση που ακολουθήσουμε την ε, γραμμή σας. Υπάρχουν και πολλές άλλες τεχνικές λεπτομέρειες, στις οποίες μπορούμε να αναφερθούμε αργότερα στη διαδικασία αυτή. Αλλά θα ήθελα να ξανατονίσω ότι θα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να υποβάλουμε τροπολογίε. Είναι αδύνατον για μένα να υποβάλω σωστέ τροπολογίε μέσα σε μία εβδομάδα, τη στιγμή που χθε έλαβα την έκθεση και δεν έχω καν το οριστικό κείμενο στα δανέζικα. Τα γερμανικά μου, δυστυχώς, δεν είναι πάρα πολύ καλά. Λίγα γερμανικά μιλάω. Ναι, μπορείτε να, μελετήσετε λίγο περισσότερο. Και ε, ε, η, έκθεση για τα βιοκτώνα σίγουρα αποτελεί καλή ευκαιρία για σας. Ε, άκουσα όμως το αίτημά σας ε, και θα μεταφέρουμε την ημερομηνία στο τέλος της εβδομάδας, 5 Μαρτίου, ε, εφόσον συμφωνεί η εισηγήτρια. Πέντε μέρες παραπάνω. Έτσι θα έχετε και στα δανέζικα το κείμενο. Ωραία. Από τους εισηγητές η Κορίν Λεπάς δεν είναι εδώ, Μισελ Λεπάς δεν είναι εδώ, Τζούλι Κέρλινγκ, όχι, απουσιάζει. Από την Επιτροπή ΙΜΚΟ, Αμάλια Σαρτόρη, επίσης δεν είναι εδώ. Ωραία Ρώση. Και η κυρία Βίλς είναι εδώ. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι πέντε μέρες αναβολής δεν επαρκούν λόγω του είδου εργασία που απαιτεί αυτό το κείμενο που είναι περίπλοκο και δύσκολο και που θα δημιουργούσε σε περίπτωση λάθους εκ μέρου μας θα δημιουργούσε λοιπόν τεράστια προβλήματα και για την δημόσια υγεία αλλά και για τους παραγωγού και τους χρήστε αυτών των ουσιών. Καταρχήν θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ βιοκτώνων και βιοκτώνων. Επειδή ακριβώς υπάρχουν κάποια βιοκτώνα τα οποία είναι σχεδόν αυλαβή και τα οποία χρησιμεύουν ε, επί παραδείγματι για να απομακρύνουμε από τα σπίτια μας τα κουνούπια και που στη συσκευασία θα πρέπει να αναφέρεται αυτή η χρήση τους και θα πρέπει και ότι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για οικιακή χρήση και υπάρχουν άλλα βιοκτώνα που τα χρησιμοποιούμε για τα κουνούπια πάντοτε για την εξαφάνισή τους που είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία υπό συγκεκριμένε ώρες και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία για παράστα και έντομα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό, συγκεκριμένε συνθήκες με κλειστά παρά, μάλλον με κλειστά παράθυρα κλπ. κλπ. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον τρει κατηγορίε αυτών των προϊόντων για την ίδια χρήση για τα κουνούπια. Το πρώτο το οποίο όπως λέγαμε είναι αυλαβές για το σπίτι αφού όλοι τέλο πάντων χρησιμοποιούμε διάφορα είδη βιοκτώνων τα οποία είναι αυλαβή. Δεύτερο είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό για να απομακρύνει να σκοτώσει τέλο πάντων τα κουνούπια από τον κήπο. Και έχουμε την έκτακτη παρέμβαση η οποία γίνεται από ειδικού για να αξιδώσουμε τέλο πάντων ολόκληρες απικίες με παράσιτα, κουνούπια κτλ. κτλ. Όπως βλέπετε λοιπόν έχουμε διαφορετική χρήση ουσιών οι οποίες παραμένουν στο περιβάλλον και που θα μπορούσαν να ήταν βλαβερές. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πάρα πολύ. Όταν μιλάμε για αμυκητοκτώνα εδώ, που είναι πάντοτε βιοκτόνα, αυτά παραμένουν στο εσωτερικό γενικά του προϊόντος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν χρόνοι μη επεξεργασίας, ώστε να είναι αυτό το προϊόν βρόσιμο. Βεβαίω το μυκητοκτόνο το οποίο πάει στο φυτό δεν το τρώμε, αλλά το μυκητοκτόνο το οποίο μπαίνει στην ε, διατροφική αλυσίδα το καταναλώνουμε. Οπότε ανεξάρτητα από την ε, επικινδυνότητα, αν εγώ τρώω ένα προϊόν το οποίο αρχικά δεν θα είναι ενδεχομένω βλαβερό, αλλά μετά από 30 μέρε θα γίνει βλαβερό, τότε εγώ θα προκαλέσω βλάβη στον εαυτό μου. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τον χρόνο εισαγωγή τέλο πάντων του βιοκτώνου στο εσωτερικό του προϊόντο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή εγώ θα μπορούσα να φάω ή όχι, τέλο πάντων φαρμάκι, αυτή είναι η δική μου επιλογή ένα άλλο θέμα. Δεν είναι όλα τα φρούτα τα ίδια. Εγώ ας πούμε θα μπορούσα να λάβω υπόψη μου ένα καρπούζι που θα μπορούσα να υποβάλω σε επεξεργασία εξωτερική με ένα αντιπαραστατικό, επειδή ξέρω ότι κανείς δεν τρώει τέλος πάντων το, τη φλούδα του καρπουζιού ή του πεπονιού. Το ίδιο και με το μήλο. Αν κάνω επεξεργασία ε, στο μήλο με διαφορετικό προϊόν το πράγμα γιατί τρώμε και τη φλούδα του μήλου. Οπότε υπάρχει ο κίνδυνος ε, δηλητηρίασης. Μετά έχουμε και για άλλα φρούτα διαφορετικές έτσι, περιπτώσεις όπου τα κατανοούμε ολόκληρα φράουλα, κεράσια, τα οποία είναι πολύ πιο έτσι ιδιαίτερα, ιδιόμορφα σε σχέση με άλλα φρούτα, γιατί κανείς τέλο πάντων δεν καθαρίζει, δεν βγάζει τα φλούδια από τα κεράσια ή από τις ε, φράουλες επειδή ας πούμε το κεράσι μαζί με τα μήλα, αλλά τώρα που έλεγα για τα κεράσια, τα κεράσια λοιπόν είναι από τα αγροτικά υγειορικά προϊόντα που υποβάλλονται σε περισσότερες χημικές επεξεργασίες και το, το τρώμε ολόκληρο. Τώρα για τους κανόνες για τη σήμανση, αν διαβάσουμε αυτό το κείμενο θα τρομάξουμε, γιατί de facto αν θα πρέπει να εφαρμόσουμε το κείμενο το οποίο φτάνει στην Επιτροπή, τότε θα κάνουμε αδύνατη την άμεση πώληση όλων των φρούτων αυτού του είδους, του δάσους, δηλαδή φράουλες, ε, κεράσια κτλ. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μεμονωμένη σήμανση για το κάθε κεράσι χωριστά σε όλες τις αγορές της Ευρώπης από τους παραγωγούς. Επειδή πολύ συχνά και ιδιαίτερα όταν είναι ε, στα πλαίσια της εποχής πολλούνται με το κιλό ε, σε τεράστιες ποσότητες. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε τη σήμανση στην ε, συσκευασία τη στιγμή που δεν υπάρχει συσκευασία, επειδή υπάρχει ένα σωρό, ε, με φράουλε, από τι οποίε παίρνει τι φράουλε ο παραγωγό και τι πουλάει. Πού θα βάλουμε λοιπόν τη σήμανση. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε και σήμανση για την άμεση πώληση που δεν προβλέπεται σε αυτό το κείμενο. Γι' αυτό ακριβώ, Πρόεδρε, ζητώ το εξή. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά για να αποφύγουμε τη δημιουργία μεγάλων προβλημάτων και στον παραγωγό αλλά και στον καταναλωτή. Οπότε ζητώ μια αναβολή πιο ουσιώδη ευρύτερη δηλαδή, για να συνεργαστούμε με, την Επιτροπή και να συντάξουμε ένα καλό κείμενο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε. Ευχαριστώ κύριε Ρώση. που μας κάνατε μία εισαγωγή στην, ε, στα φρούτα. Υπάρχει η φλούδα των καρπουζιών και η φλούδα των, ε, των φραουλών. Ε, η κυρία Κλάστα απαντήσει η κυρία Αντώνια Παβανόβα και Σαμπίνε Βίλς. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω εκ μέρους κυρίου Ναβάσου, η οποία ζητάει συγγνώμη που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα εδώ. Πιστεύει ότι η συγγήτρια έχει ε, εκπονήσει μια πολύ καλή έκθεση. Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο και όπως ανέφερε δεν μπόρεσε να επισέλθει σε λεπτομέρειες και έλαβε την έκθεση μόνο αγγλικά και γαλλικά και μάλιστα πολύ αργά. Γι' αυτό το λόγο ε, συμφωνούμε να παραταθεί προθεσμία για τις τροπολογίες και συμφωνούν ότι μία εβδομάδα δεν αρκεί ε, δεδομένου ότι το θέμα είναι πολύ τεχνικό, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Στο παρόν στάδιο λοιπόν η έκθεση ε, δημιουργεί ορισμένα σχόλια από εμά. Καταρχήν, η κ. Λεπάζ χαιρετίζει ορισμένε τροπολογίε επειδή βελτιώνουν την πρόταση επιτροπή, για παράδειγμα, όσον αφορά την προστασία, τα είδα τα νέε διατάξει και επίση συμφωνεί ε, ω προ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, επίση συμφωνεί με την τροπολογία τη ηγήτρια 10 για την προστασία ε, τη υγεία των ζώων και των ανθρώπων κατόπιν η έκθεση δεν ε, ασχολείται με βασικές προκλήσεις επιτροπής. Όσον αφορά το 5, η διευκρίνηση αυτού του άρθρου είναι κάτι πολύ καλό, αλλά η έκθεση ακόμη επιτρέπει ε, σε ορισμένες τοξικές ουσίες ε, να, υπάρχουν στην αγορά. Επίσης, η κυρία Λεπάζ ανησυχεί όσον αφορά την παρέκκληση από τα αποκλειστικά κριτήρια του άρθρου 5. Θα ήθελε να ζητήσει στην εισηγήτρια και στην Επιτροπή κατά πόσο το άρθρο 45 δεν θα αρκούσε ε, όταν ε, υπάρχουν προβλήματα εκτάκτου ανάγκης. Γι' αυτό τον λόγο η κυρία Λεπάζ ε, στην Επιτροπή ζήτησε μια τροπολογία για να απαλληφθεί αυτή η παρέκκληση στο άρθρο 5. Όσον αφορά την προσέγγιση μικρή επικινδυνότητα, συμφωνεί, αλλά θα ήθελε καλύτερο ορισμό των προϊόντων που δεν συνιστούν μεγάλο κίνδυνο, για παράδειγμα. Η απουσία έκθεση δεν είναι επαρκή λόγο ε, για ε, να θεωρηθεί όταν, ε, ότι ένα προϊόν δεν έχει μεγάλο κίνδυνο. Τώρα, η προσέγγιση τη εισηγήτρια είναι να δώσει κεντρική αδειοδότηση για κάθε ε, η κυρία λοπάζου δεν έχει Η... Θα πρέπει αυτό το θέμα να συζητηθεί λοιπόν όσον αφορά ε, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Ε, θα, η κυρία Λεπάζ θα ήθελε τα οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανεκατασταθούν με ε, τις, ε, τα προγράμματα αξιολόγηση των παρασιτοκτόνων της ε, Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Δεν έχει πιστεί ότι αυτό το πρόγραμμα ταποκρίνεται στα, στους κανόνες τους περιβαλλοντικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τη διαφάνεια και το θέμα των υλικών, Η κυρία Λεπάζ ε, λυπάται που δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία δημοσιοποιημένα όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Όσον αφορά τις πληροφορίες λοιπόν επί της ουσίας, ε, δεν υπάρχουν, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και οι στατιστικές θα έπρεπε να δημοσιοποιούνται και να ενημερώνονται τακτικά. Κυρίως ζητάει να υπάρχει μια έκθεση για τι τις επιπτώσεις των νανοηλικών και θα καταθέσει σχετικά μια τροπολογία. Και όπως σας είπα, ίσως η καλύτερη ιδέα θα ήταν να υπάρχει συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών, ώστε να μπορέσουν να σχολιάσουν περισσότερο το θέμα ε, και να κάνουν σχετικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Σαμπίνε Βίλς. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι σκιώδη εισηγήτρια για την ΚΟΕ. Η κυρία Κλάς έχει εκπονήσει μια έκθεση πολύ φιλική προς τη βιομηχανία κατά τη γνώμη μου. Η αναθεώρηση του κανονισμού για την αδειοδότηση των βιοκτώνων δεν, ε, δεν πληρεί τα πρότυπα του, της οδηγίας για τα παρασιτοκτώνα, για τα φυτοφάρμακα. Ε, έχει περιοριστεί εκεί βέβαια το πεδίο εφαρμογής, ε, ενώ τα βιοκτώνα χρησιμοποιούνται από όλους τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα προβληματικό στην πρόταση κανονισμού για τα βιοκτώνα είναι οι προϋποθέσεις αδειοδότησης προϊόντων χαμηλής επικινδυνότητας. Θα ήθελα να στηρίξω αυτό που ήδη υπόθηκε. Ε, ότι η αδειοδότηση των ε, βιοκτώνων ε, στα οποία δεν εκτίθεται ο κόσμος εδώ θα ήθελα να πω ότι τα βιοκτώνα χρησιμοποιούνται από όλους, ιδιαίτερα από ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι έγκυοι και τα παιδιά. Η αποφυγή τους στην καθημερινή ζωή είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει και συγκεκριμένα προϊόντα με τη λεγόμενη χαμηλή επικίνδυνοτητα που ε, έχουν λάβει άδεια μόνο σε ένα κράτο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού και αυτό το θεωρώ σημαντικό πρόβλημα. Όσον αφορά την ε, ευρωπαϊκή αδειοδότηση βιοκτώνων, εγώ πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μην επιτρέψουν τη χρήση ε, κάποιων βιοκτώνων στη χώρα τους. Ε, είναι πολύ διαφορετική η χρήση των βιοκτώνων που γίνεται από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Για παράδειγμα, ε, στο σπίτι ή η δημόσια χρήση εντομοκτώνων γίνεται με διαφορετικό τρόπο και είναι πολύ δύσκολο η επιστημονικές έρευνες να ορίσουν τη χρήση που γίνεται από, το, από τους ανθρώπους. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, όπου η χρήση γίνεται από ε, επαγγελματίες είναι πολύ πιο εύκολο να ορίσει κανείς πώς γίνεται η χρήση. Όσον αφορά την απαγόρευση συγκεκριμένων ε, ουσιών, όπως για παράδειγμα τα ανανοήλικα, αυτά υπάρχουν στα μπιπερό, στην οδοντόκρεμα, σε συσκευασίες τροφίμων και είναι πολύ δύσκολο τόσο βραχυπρόθεσμα μετά την υποβολή της έκθεσης να συζητήσουμε όλες τις διάφορες ε, πτυχές, ε, τις συνέπειες ε, στους καταναλωτές. Υπάρχει ανάγκη για περισσότερη εξέταση. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό που υπόθηκε να επεκταθεί η προθεσμία για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Κάρλ θα ήθελα καταρχήν να υποστηρίξω το αίτημα του Νάνσε για να παραταθεί η προθεσμία για την κατάρτιση τροπολογιών. Χρειάζεται σε ένα περίπλοκο θέμα όπως αυτό. Θα ήθελα να αναφέρω τα θετικά στοιχεία που βρήκα στην έκθεσή σας, κυρίως για τη βελτίωση του άρθρου 5. Η Επιτροπή έκανε ένα λάθος μεγάλο να μην περιληφθούν τα PPT, τα PPT και αυτές οι ουσίες στο κατάλογο. Συνεπώς αυτή είναι μια βελτίωση. Επίσης είμαι σε ευτυχή ω συνήθω να βλέπω και τα νάνο στοιχεία και η παραδεκτή μορφή. Χαίρομαι που τα αναφέρετε. Είναι ένα σημαντικό θέμα ε, το οποίο δεν έχει καμία γνώση ο καταναλωτής. Δεν συμφωνώ με σας να απαλείψουμε εντελώ τις ευθύνε για τα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες, ε, τα έθη και τα έθιμα είναι διαφορετικά, υπάρχουν ορισμένε ε, συμφωνίες που γίνονται μεμονωμένες, γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και θα ήθελα να γνωρίζω αν ε, ο οργανισμός των χημικών ουσιών έχει τη διοικητική ικανότητα να αντιμετωπίσει το επιπλέον βάρος που υπάρχει, λαμβάνοντας υπόψη την πίεση που ήδη αντιμετωπίζει. Επίσης θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερο περιοριστικά κριτήρια εδώ. Για παράδειγμα, αν δούμε το άρθρο 5.2β. Εάν θεωρηθεί ότι πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με την εμπειρία μου και αφού συνάντησα κυρίω ε, του υπεύθυνου τη περιοχή τη Στοχόλμη για τα νοσοκομεία, την υγιεινή, ε, μου ανέφερε ότι πολύ συχνά ακόμα και στα νοσοκομεία είναι καλύτερα να χρησιμοποιεί κανεί απλά το ενόπνευμα για να καθαρίσει επιφάνειε. Ε, και ε, εάν έχετε μαζική χρήση On Διοκτώνα βλέπουμε ότι ε, ε μερικές φορές ε, χρησιμοποιούνται χωρίς να είναι απαραίτητα. Γι' αυτό περιορίζεται η επίδρασή τους. Γι' αυτό ε, πρέπει νομίζω να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση των διοκτώνων. Επίσης, δεν συμφωνώ όταν λέτε υποσυνήθεις ε, συνθήκες χρήσης. Περισσότερα από το 50% των ετησίων εκκλήσεων τοξινών είναι όταν υπάρχει μια διαταραχή στο σύστημα. Γι' αυτό θα ήθελα να υπάρχει εγγύηση για πιο σωστή χρήση. Διότι όταν έχετε κλειστά συστήματα ή ε, πολλοί πολύ αποτελεσματικά συστήματα καθαρισμού, όταν υπάρχει διακοπή μια ώρα στο σύστημα, τότε μπορεί να ελευθερωθούν πάρα, πολλά, πάρα πολλές ουσίες περισσότερες από ό,τι έχουν σε ένα χρόνο. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν και εδώ περιορισμοί. Τέλος, υπάρχουν εγκαταστάσεις ε, καθαρισμού των υδάτων. Νομίζω βιολογικού καθαρισμού των υδάτων. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, διότι αν δεν έχουμε καλούς βιολογικούς σταθμούς και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα επιπλέον κριτήριο για να περιοριστούν αυτέ τι ουσίε. Και επίσης και η αντίσταση στα αντιβιωτικά. Βλέπετε ότι πολλά ε, ε, για πολλά προϊόντα οι καταναλωτές θεωρούν ότι δεν είναι επικίνδυνα. Θα, πω να σας, θα σας έλεγα μάλιστα ότι είναι πιο ασφαλές να έχω βρώμικα χέρια τα οποία είναι γεμάτα βακτηρίδια διότι ε, υπάρχει ανοσία αν θέλετε. Εάν έχετε εντελώς ε, αποστηρωμένα ε, χέρια, τότε έχετε μεγαλύτερους κινδύνους. Λοιπόν, δεν πρέπει να φοβόμαστε συνέχεια. Επίση, για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. δεν ξέρω τι θέλουν οι φιλελεύθεροι. Οι μικρομεσαίε συχνά δεν γνωρίζουν πολύ καλά ε, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποια είναι τα ωφέλη. Δεν έχουν αρκετές πληροφορίε. Οι περιορισμοί του βοηθούν μερικέ φορέ και άλλε φορέ του κάνουν κακό. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε πάλι ένα συμβασμό με τι μικρομεσαίε. Διότι οι κανονισμοί ε, για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στι μικρέ ουσίε μερικέ φορέ είναι καλοί, άλλε φορέ είναι επιβλαβεί. Ευχαριστώ. Επίσης υπάρχει κάποιος άλλος στους Γεια, Άνια Βάισκαβα. Ωραία, η Άνια Βάισπερκερ. Πρόεδρε, κυρία εισηγήτρια, καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ε, καλή αυτή έκθεση. Βρίσκεται πολύ πλήρης, πηγαίνει προς την κατεύθυνση Κάποιες παρατηρήσεις έχω, θα ήθελα κάποια πράγματα να τα επιβεβαιώσω και έχω και κάποιες ερωτήσεις. Το πρώτο θέμα είναι η κοινοτική αδειοδότηση. Σύμφωνα με την ε, υπάρχουσα οδηγία θα πρέπει όλα τα βιοκτώνα να εγκρίνονται από τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν προτείνει πέρα από την ε, αδειοδότηση των ε, κρατών μελών να υπάρχει και ευρωπαϊκή μόνο για τα προϊόντα όμως χαμηλής επικινδυνότητας και προϊόντα που περι... και μόνο προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες. Η έκθεση αυτή πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση, όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι μισό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Χαίρομαι που η συγγήτρια τολμά ε, το βήμα προς την πλήρη εναρμόνιση και που στο σχέδιο έκθεσης ε, προτείνει την ε, ε, κεντρική αδειοδότηση για όλες τις ουσίες. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η Κομισιόν στην μελέτη επιπτώσεων γράφει ότι η κοινοτική αδειοδότηση θα ήταν πιο αποτελεσματική. Γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτήν την οδό και και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να γίνεται κεντρικά η αδειοδότηση για όλες τις ουσίες. Κάποια θέματα τα γνωρίζουμε από τον κανονισμό για τα φυτοφάρμακα. Θα ήθελα να ξέρω τι έχει γίνει κατά τις πρώτες συζητήσεις στο Συμβούλιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα και πιστεύω ότι θα πρέπει να το τονίσει το Κοινοβούλιο και ενδεχομένω να έχουν και όλες οι πολιτικές ομάδες σε την ίδια γνώμη. Βρίσκω επίσης πολύ καλή τη λύση στο σχέδιο της ε, έκθεσης ε, να μπορεί να γίνουν ε, οι δοκιμές σε ένα κράτος μέλος, διότι ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σημαντικό να μην πρέπει απαραίτητα να συνεργάζονται με το Ελσίνκι, αλλά να έχουν και συνομιλητές σε εθνικό επίπεδο. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά τα νανοηλικά και ιδιαίτερα τον προτινόμενο ορισμό. Πέρσι τον Απρίλιο στο Στρασβούργο υιοθετήσαμε ψήφισμα για τα νανοηλικά, όπου διαπιστώσαμε ότι τα νανοηλικά ε, ε, προσφέρουν πολλές ε, δυνατότητες στον ε, τομέα ε, της βιομηχανίας, ε, στην κατασκευή αυτοκινήτων, στην οπτική, στα φάρμακα. Δεν θα πρέπει να κλείσουμε τα μάτια σε αυτές τις δυνατότητες ανάπτυξης και έρευνας. Θα πρέπει όμως να χειριστούμε τα θέματα αυτά και με την απαραίτητη ευαισθησία και προσοχή. Εδώ, Κρίστα, έχει συμπεριλάβει ορισμό για τα νανοηλικά πιστεύω ότι είναι και ένας από τους πρώτους ορισμούς νανοηλικών που συναντούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ορίσουμε τα νανοηλικά στην υπάρχουσα νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε αν ο ορισμός αυτός ε, ισχύει μόνο στην περίπτωση των διοκτώνων ή αν θα πρέπει ε, να... Ε, ή αν θα μπορούμε να τον εφαρμόσουμε και σε άλλους τομείς. Θα ήθελα λοιπόν πολύ να το εξετάσω αυτό σε συνεργασία μαζί σου. Η τρίτη μου παρατήρηση αφορά την αδειοδότηση των προϊόντων διοκτώνων Στο μέλλον Ε, τα προϊόντα θα μπορούν να τυχαίνουν μεταχείριση από βιοκτώνα μόνο εφόσον τα βιοκτώνα αυτά έχουν εγκριθεί εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει και για εισαγόμενα προϊόντα. Όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή, θα μπορούσε να πει κανεί ότι κάτι τέτοιο πηγαίνει προ σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω όμω ότι η υποχρέωση Αυτή θα έχει ιδιαίτερες συνέπειες ε, για την εισαγωγή χημικών ουσιών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τίθεται το ερώτημα πώς, ε, θα, πώς μπορεί να ελεγχθεί αυτό. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και τη γνώμη της Κομισιόν. Διότι όταν μιλάμε για προϊόντα βιοκτώνων, είναι σημαντικός ο έλεγχος ε, και θα πρέπει να, ο έλεγχος να επικεντρώνεται κυρίως στην χημική δραστική ουσία. Έχουμε τα κριτήρια από τον ε, τομέα των φυτοφαρμάκων. Ε, είναι αυστηρά τα κριτήρια αυτά γιατί θα πρέπει επιπλέον να γίνεται ειδική αδειοδότηση για τα βιοκτώνα και τι θα, πώς θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος στα εισαγόμενα προϊόντα. Πρώτη τελευταία παρατήρηση, τα τέλη. Σημαντικό είναι να υπάρχει εναρμόνιση όσον αφορά το ύψος των τελών. Ε, πιστεύω ότι τα ετήσια τέλη για τα οποία δεν λαμβάνει και κανείς τίποτα, είναι προβληματικά ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό συμφωνώ με τη διαγραφή ε, των τελών αυτών και επίσης όσον αφορά την αδειοδότηση των προϊόντων χαμηλής ε, Ίσως θα, μπο... θα έπρεπε στον τομέα αυτών και υπάρχει σαφής ορισμός ε, σχετικά με το τι είναι χαμηλή επικοινωνότητα, Ίσως θα έπρεπε εδώ να εισάγουμε ε, ένα σύστημα επισήμανσης ώστε ο καταναλωτής να λαμβάνει τα σχετικά σχετικές πληροφορίες, να γνωρίζει δηλαδή ότι ε, χρησιμοποιεί ένα ασφαλές προϊόν. Έτσι μπορεί να ε, γίνει σχετική διάκριση και ε, να παρέχουμε σωστό επίπεδο προστασίας. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση και προσλέπω στην καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τον λόγο στην Κομισιόν, τον κύριο Πολ Σπέτ. Προτού να ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να απαντήσει. Κύριε Σπέτ. Yeah. thanks, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ την κυρία Κλάς για τη σκληρή δουλειά που έκανε σχετικά με την έκθεση η οποία είναι επικοδομητική συμβολή για να προχωρήσουμε όσον αφορά την αναθεώρηση ε, στο τομέα των διοκτώνων. Ορισμένα θέματα ε, τα χαιρετίζει η Επιτροπή Πρώτα απ' όλα η προσθήκη των περιβαλλοντικών κριτηρίων στο άρθρο με τις εξαιρέσεις σύμφωνα με τη θέση την οποία έχει παρουσιάσει παρουσίαση Κομισιόν στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Δεκεμβρίου δεχόμαστε το PPT, PPT, WOP, την αναθεώρηση όλων αυτών. Δεύτερο θέμα το οποίο είναι αποδεκτό από μας είναι η ειδική μνήμα στην ανάγκη να γίνεται έλεγχο στα θέματα της νανοτεχνολογίας. Παρά το γεγονός ότι αυτό θα γινόταν βεβαίω στην πράξη, αλλά καλύτερα να το καταστήσουμε σαφέστερο. Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε παρόλα αυτά την ανάγκη που ανέφερε και η vice Κάμπρελ, να δούμε με προσοχή τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται. Και από ό,τι καταλάβαμε, αυτό είναι ο ορισμός ε, που αφορά τα νέα τρόφιμα. Και η Επιτροπή αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βρει ε, ε, μία, έναν γενικό τρορισμό για τα προϊόντα της νανοτεχνολογίας. Και πιθανόν θα μπορούσαμε στην πρώτη ανάγνωση ε, να το προσθέσουμε. Επίσης ένα άλλο επικοδομητικό σημείο είναι οι τροπολογίες για ε, την διάταξη που αφορά τα προϊόντα επεξεργασίας και το διαχωρισμό μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων. Και αυτό πλουστεύει τα πράγματα και εκεί νομίζω το Συμβούλιο συμφωνεί. Επίσης ε, παραδεχόμαστε ότι οι τροπολογίες για τη σήμανση και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε με προσοχή πώ θα λειτουργήσει στην πράξη. Η κυρία Κλά αναφέρθηκε στου εξωτερικού παράγοντε που το καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Απλά σημειώνουμε ότι ορισμένα από τα ε, πρόσφατα προβλήματα που είχαμε με τα βιοκτώνα αφορούσαν περισσότερο ε, τις εσωτερικές επιπτώσεις όπως ε, εξανθήματα για παράδειγμα. Just a word of caution on that. Ε, δηλαδή που, που έρχονται από του καναπέδε. Ε, η τροπολογία να για την ενημέρωση του κοινού το χαιρετίζει η Κομισιόν, έχει δίκιο η κυρία Κλάσε που το υπογραμμίζει. Πρόκειται ένα σημαντικό σημείο των θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των βιοκτώνων, αλλά μπορούμε να ερωτηθούμε κατά πόσον αυτή η ιδέα της αηφόρου χρήσης των βιοκτώνων ε, μπορεί να τοποθετηθεί στην οδηγία ή την αγορά. Η Επιτροπή το μελετάει αυτό το θέμα και δεν ξέρω αν είναι αυτό το σωστό νομικό κείμενο. Είναι προσυζήτηση το θέμα. Τώρα ως προς τα σημεία ε, που παρουσιάζουν δυσκολίες για την Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι υπάρχει συνδυασμός ε, μεταξύ επιπλέον βάρου εργασία και λιγότερου χρόνου για την ΕΚΑ στην έκθεση. Αυτό έχει ορισμένε επιπτώσει, φυσικά αναπόφευκτα Κυρίω η τροπολογία 67 που αναφέρεται σε τροπολογία από 9 μήνε ή 3. Ένα παράδειγμα που θα παρουσιάσει πρόβλημα. Θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή, ώστε ο οργανισμό να μπορεί με αηφόρο τρόπο να το αντιμετωπίσει χωρί να δημιουργήσει προβλήματα ε, στο, στην εργασία του. Ε, Ορισμένα άλλα μέλη ανέφεραν ότι ε, ο συγκεντρωτικός, η συγκεντρωτική αντιμετώπιση είναι ένα ε, ε, σωστό είναι πρόβλημα όπως έδειξε η εκτίμηση επιπτώσεων πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να βρούμε πάλι τη χρυσή τομή. Δεν ξέρουμε πόσα προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά. Μπορεί να είναι 10.000 προϊόντα, πάρα πολλά είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να διαχειριστεί, δηλαδή ο οργανισμός μπορεί να το διαχειριστεί. Αμφιβάλλουμε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βρεθεί εδώ κάποιος συμβιβασμό. Ένα άλλο σημαντικό θέμα και, σε και επικεντρώνονται πολλές τροπολογιστικές κλάσεις πάνω αυτό το θέμα είναι η ισορροπία μεταξύ ε, των ομάδων βιομηχανίας που βρίσκονται στο πρόγραμμα αναθεώρησης και έχουν τα χρήματα και οι ομάδες που βρίσκονται εκτός ονομάζονται free writers Σε ορισμένε περιπτώσει όμω ε, είναι μικρομεσαίε ε, που έχουν πολύ μικρό μερίδιο τη αγορά. Και πιστεύουμε ότι νόμιμα μπορούν ε, να βρουν μια θέση στην αγορά σε ένα δεύτερο στάδιο. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να μην τους βγάλουμε έξω από την αγορά, αλλά να έχουν την ευκαιρία να βρουν μια θέση στην αγορά. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε περαιτέρω. Είμαστε ε, ανοιχτοί ε, σε μερικές ιδέες ε, της σχέσης κλάσης ως προς την εφαρμογή του άρθρου 86, αλλά θα πρέπει να μην δημιουργούνται μονοπόλια και να μπορούν και άλλες εταιρείες να βρουν μια θέση στην αγορά και να εμπορεύονται. Ορισμένες μικροπαρατηρήσεις τώρα όσον αφορά η, διαγραφή της ετήσιας συνδρομής. Ε, η ιδέα της ετήσιας συνδρομής ήταν να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχει κατανομή των δαπανών. Αντί να πληρώνει κανείς ένα μεγάλο ποσό στην αρχή, να πληρώνει μικρά ποσά σταδιακά. Και να υπάρχει κατανομή των δαπανών. Επίσης, σημειώνουμε ότι υπάρχουν πολλές τροπολογίες για την ιδέα ε, των ε, συμπληρωματικών ε, ομοίων προϊόντων. Αυτή είναι η εμπορική πρακτική, αλλά δεν νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να περιληφθούν σε ένα νομικό κείμενο, Διότι γίνεται πολύ περίπλοκο το επίσημο κείμενο. Τέλος, τρεις παρατηρήσεις σχετικά με τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Ο κύριος Γιόργενσεν, ναι, η Επιτροπή πράγματι είναι ανοιχτή όσον αφορά τις περισσότερη δουλειά να γίνει για τα προϊόντα χαμηλού κινδύνου. Ε, πρέπει τα προϊόντα να είναι αξιόπιστα, πιθανόν λειτουργικά, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε εδώ το θέμα. Και με τα χαράς ε, θα καταβάλουμε προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά, ένα ερώτημα για τις παρεκκλήσεις από, όσον αφορά τα κριτήρια αποκλεισμού και ε, σε σχέση με το άρθρο 45. Πιστεύουμε ότι το άρθρο 45 έχει ως αντικείμενο την καταπερίπτωση εξέταση και για μικρή διάρκεια. Ε, όσον αφορά τις εξαιρέσεις και τις παρεκκλήσεις είναι ε, ορισμένα παρασιτοκτόνα ή όταν υπάρχει δηλητηρίαση ε, από το δηλητήριο για τα ποντίκια για παράδειγμα πριν από ένα 1,5 χρόνο το είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα εδώ δεν είναι παρέκκληση κατά περίπτωση αλλά έχει, θα το, δέχεστε το δηλητήριο για τα ποντίκια, και το ποντικοκτόνο ή όχι. Πρέπει ε, το αποτέλεσμα είναι πιο προβλέψιμο. Η τελευταία ερώτηση ήταν της κυρίας Βάις Γκέρμπερ, πώς θα εφαρμόσουμε ε, τα προϊόντα τα οποία ε, έχουν είναι αντικείμενο επεξεργασία. Η παρούσα κατάσταση δεν είναι αποδεκτή, διότι είχαμε προϊόντα στην υγεία από αυτά τα προϊόντα και υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός όσον αφορά τους κοινοτικού παραγωγούς. Βεβαίως θα πρέπει να βρούμε μια πρακτική λύση, όχι να έχουμε τους τελωνιακούς που θα ελέγχουν το κάθε προϊόν, όχι βέβαια. Γι' αυτό ε, υπάρχουν ορισμένες διατάξεις που έχουν σχέση με τη σήμανση, μια προσπάθεια δηλαδή να διευκολύνουμε τις ε, εποπτικές αρχές ώστε να βρουν τα προϊόντα τα οποία πιθανόν θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή. Η εισηγήτρια έχει το λόγο. Κρίστα Κλάς. να αναφερθώ και στο χρονοδιάγραμμα. Έχω εδώ πέρα την πρόταση να ε, μεταθέσουμε την προθεσμία για τις τροπολογίες 5η 11 Μαρτίου, την 5η του Στρασβούργου. Ε, έτσι κινδυνεύουμε όμως 6-7 Απριλίου να μην έχουμε τις ε, μεταφράσεις. Μπορούμε όμως βέβαια να το δοκιμάσουμε διότι αυτό είναι επιθυμία από πολλές πλευρές. Ε, θα ήθελα επίσης πριν σας δώσω το λόγο να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών από την ε, εκλογική περιφέρεια της Ντάγμα Ροτ Πέρεντε. Αναφερόμαστε σε μια πρόταση που αφορά τα βιοκτώνα όπου θέλουμε ε, να εισάγουμε προληπτικούς κανόνες. Η συγκήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέρφους που ζήτησαν το λόγο. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας συζήτησης η οποία είναι απαραίτητη εδώ στην νομοθετική διαδικασία και ελπίζω ότι θα υπάρξουν και μελλοντικέ συζητήσει. Η συζήτηση η σημερινή ήδη έδειξε πόσο διαφορετική είναι η προσέγγιση των διαφόρων προς τα βιοκτώνα. Ως προς ε, το χρονοδιάγραμμα, κύριε Πρόεδρε, εγώ προσωπικά δεν έχω πρόβλημα με τις 11 ε, Μαρτίου. Επανειλημμένα έχουμε προβλήματα με τη μετάφραση. Ε, όλο και κάποιος λέει ότι δεν όλο και κάποιο λέει ότι α, δεν έχω τι τροπολογίε στι χώρε μου, ε, ε, στη γλώσσα μου, συγγνώμη. Ε, ε, να πούμε λοιπόν ήδη τώρα ότι όποιο υποβάλλει τώρα τι τροπολογίε του θα προλάβει να τι δει και μεταφρασμένε. Εάν δηλαδή αργήσετε να υποβάλλετε τι τροπολογίε σα μπορεί να μην μεταφραστούν εγκαίρω. Εγώ πάντως συμφωνώ με τι 11 Μαρτίου, ελπίζω όμω ότι θα μπορέσουμε ε, όλοι να υποβάλουμε τι τις τροπολογίες μας, ε, ώστε να έχουμε εγκαίρω και τη μετάφραση. Ε, έχω γράψει εδώ προσεκτικά τις παρατηρήσει των συναδέρφων. Παρακαλώ μην περιμένετε απάντηση σε κάθε ερώτηση από μένα τώρα. Ε, και σε κάθε εκκλησία ήταν Γιώργενσεν. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά για τα φυτοφάρμακα και πιστεύω ότι γνωρίζουμε τη σημασία των παρασιτοκτόνων και των βιοκτόνων και στην συζήτηση σίγουρα θα ε, εισάγουμε τα συμπεράσματα που είναι σημαντικά για μας. Ε, τα βιοκτώνα θα πρέπει να βοηθούν τους ανθρώπους, όχι να τους λάπτουν. Ε, αυτή η προσέγγιση ε, νομίζω ότι είναι κοινή, έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Και νομίζω ότι το αναγνωρίζουμε αυτό και οι δύο. Όσον αφορά την κατάργηση των παρεκκλήσεων, η Κομισιόν τις οποίες τη θέση συμμερίζομαι, ε, πιστεύει ότι είναι απαραίτητες οι παρεκκλήσεις για ε, τα βιοκτώνα. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όταν δεν υπάρχει κάποια ουσία υποκατάστατο, τότε θα πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο βιοκτόνο. Γι' αυτό παραμένουν οι μεταβλητές ε, και άλλες ε, πολιτικές ομάδες ε, έχουν συζητήσει το θέμα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τις παρεκκλήσεις. Η δημιουργία άλλης νομικής βάσης, αυτό θα πρέπει να συζητηθεί. Έχουμε τώρα τη νομική βάση της εσωτερικής αγοράς, η οποία κατά τη γνώμη μου αρκεί Οτιδήποτε άλλο θα ε, δυσκολέψει τις εργασίες, ε, θα το συζητήσουμε όμως. Όσον αφορά την ε, δυνατότητα ανησυχίας κατά την αδειοδότηση, γνωρίζω την δανέζικη προσέγγιση. Τα κράτη-μέλη δηλαδή να έχουν δικαίωμα ανησυχία κατά την, κοινωνική την κοινοτική αδειοδότηση. Συγγνώμη. Έχουμε λοιπόν μία κοινή αγορά Θέλουμε να μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, θέλουμε όμως και τις εθνικές ε, παρεκκλήσεις. Ως προς τα παραστοκτόνα υπάρχουν ε, οι κλιματικές διαφορές. Και ε, ναι, το αν, έχουμε, το αν φυτρώνουν κεράσια ή δημητριακά ή μιμήλα, αυτό εξαρτάται από τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. Στα Παρασιτοκτόνα λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρχουν ε, διαφορές. Ε, για τα βιοκτόνα εγώ το αμφισβητώ αυτό διότι θέλουμε να αγοράζουμε για παράδειγμα και στην Ιταλία όταν πηγαίνουμε διακοπές το ίδιο προϊόν που βρίσκουμε στη Γερμανία. Ας ε, το συζητήσουμε όμως για να βρούμε μια κοινή προσέγγιση. Ο συνάδελφος Ρώση μίλησε και έτσι νιώθουμε και τις διαφορές που υπάρχουν ε, και στα παρασιτοκτόνα είχαμε κολλήσει. Δεν μιλάμε εδώ ε, για ε, επικόλληση ετικέτας στα κεράσια. Αυτό το ρυθμίσαμε στον κανονισμό για τα παρασιτοκτόνα που μιλήσαμε για μέγιστα όρια υπολοιμάτων. Εδώ δεν ε, κάνουμε το ίδιο. Πέφτουμε πολύ εύκολα στην παλιά συζήτηση ε, της προσέγγισης ε, που βασίζεται στον κίνδυνο, την οποία εγκαταλείψαμε και στα πλαίσια των παρεστοκτώνων. Ως προς τους επαγγελματίες χρήστες, τους έχω συμπεριλάβει ε, αυτό το λέτε και εσείς, υπάρχουν διάφορα προϊόντα τα οποία ε, ε, τυχαίνουν διαφορετικής χρήσης. Όταν όμως στη δουλειά μου κάνω κάτι, έχω ευθύνη για άλλους, έχω εκπαίδευση για να κάνω τη δουλειά μου αυτή, θα πρέπει να γνωρίζω τι κάνω και γι' αυτό οι επαγγελματίες χρήστες, οι υπεύθυνοι υγιεινή σε ένα νοσοκομείο για παράδειγμα θα πρέπει να γνωρίζουν τι προϊόν χρησιμοποιούν και πώς. Η νοικοκυρά που χρησιμοποιεί εντομοκτόνο κατά των κουνουπιών. Θα πρέπει να διαβάσει την ετικέτα και ενδεχομένως να ενημερωθεί από τον πολιτή. Θα πρέπει να, γίνουν, ε, να γίνει διάκριση εδώ. Κυρία Παρανόβα, αναφερθήκατε στην ε, μεταφορά της προθεσμίας. Συμφωνήσαμε σχετικά με το θέμα αυτό ανησυχία για τις ε, παρεκκλήσεις. Ε, αυτό ήδη το είπα στον Νταν Γιώργενσεν. Θα πρέπει να φροντίσουμε και την εσωτερική αγορά όταν μιλάμε για κεντρική αδειοδότηση. Η συνάδελφος Βίλς είπε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα απαγόρευσης μιας ουσίας και αυτό έχει να κάνει με την εναρμόνιση στην ενιαία αγορά. Προς τον ε, συνάδελφο Σλίτερ που δυστυχώς ε, λείπει τώρα, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον είναι γνωστό ότι ε, δεν έχουν τόσο καλή ανοσία όσο τα παιδιά που παίζουν με στη λάσπη Θα πρέπει να το φροντίσουμε το θέμα αυτό στην ε, κοινωνία μας, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι όσο λιγότερο πλένουν τα χέρια μου τόσο, πιο, τόσο καλύτερη ανοσία έχω. Θα πρέπει να φροντίσουμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Η συνάδελφος Βάις Γκέρμπερ αναφέρθηκε στα νανοηλικά. Η κυρία Ροτμπέρεν ξέρει περί τίνος μιλάω. Έχω πάρει τον ορισμό από τον, ε, τον κανονισμό για τα καινοτόμα τρόφιμα, για τα novel foods. Θέλουμε να βρούμε έναν ορισμό που να ταιριάζει σε όλους τους τομείς. Θα πρέπει να ε, ακολουθήσουμε εδώ την ε, έρευνα, την καινοτομία και να δούμε τι ακριβώς είναι απαραίτητο. Πιστεύω ότι πολύ σωστά αντιμετωπίζουμε εδώ τα νανοηλικά και ε, ο ορισμός, ε, και το ξέρει η δάγμα Ροτ θα είναι ο τελικός οριστικός, ε, αλλά σίγουρα αποτελεί μια καλή προσέγγιση το να λάβουμε υπόψη μας τα νανοηλικά. Άνια Βάισκερπερ αναφέρθηκε ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και στο μέλλον θα έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με το ε, κείμενό μου, να πούνε ότι έχω ένα προϊόν το οποίο θέλω να διαθέσω μόνο στην αγορά της Γερμανίας. Μπορώ λοιπόν να πάω στις εθνικές αρχές και να λάβω εθνική αδειοδότηση. Από εκεί και πέρα όμως ε, θα πρέπει να είναι δυνατόν για τι επιχειρήσεις που θέλουν να κινηθούν στην εσωτερική αγορά να πάνε κατευθείαν στην ECHA και να πούνε ότι όφελο να διαθέσω το προϊόν μου στην ευρωπαϊκή αγορά και γι' αυτό έχουμε την προσέγγιση της ε, κοινοτική αδειοδότηση. Η ECHA θα πρέπει να μπορεί να αναθέσει σε ένα κράτος εισηγητή τις ε, βασικές δοκιμές, ε, αλλά μέσω της υπηρεσίας αυτής θα υπάρξει η δικτύωση. Ε, και θα υπάρχει η ασφάλεια όσον αφορά το αποτέλεσμα των ερευνών. Πιστεύω ότι αυτό διασφαλίζεται καλύτερα εάν έχουμε αυτό το δίκτυο μέσω της ECHA. η εκκρεμότητα, η ερώτηση προς την Κομισιόν, τι θα την οποία θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω. Όσον αφορά την επισήμανση, εγώ δεν έχω φτάσει σε οριστικό συμπέρασμα. Σημαντικό είναι ένα βιοκτόνο προϊόν, το οποίο αποτελείται από διάφορες δραστικές ουσίες, οι οποίες κάθε τόσα χρόνια θα πρέπει να ελέγχονται. Ε, όλες αυτές οι δραστικές ουσίες συνδυάζονται λοιπόν σε ένα προϊόν. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τις δραστικές ουσίες ε, ή θα πρέπει να εξετάσουμε το σύνολο του προϊόντος. Ε, ας ζητήσουμε τη συμβουλή των επιστημόνων ε, είμαι ανοιχτή στη συζήτηση αυτή και στο μέλλον πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που είχαμε το χρόνο να συζητήσουμε τόση ώρα την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κλάς για τις ε, προσπάθειές σας σε αυτό το ευρύ θέμα. Ε, ημερομηνία, ε, προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 11 Μαρτίου το μεσημέρι και να σας αναφέρω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το νέο σύστημα για την υποβολή των τροπολογιών. Φτάνουμε στο σημείο 16 της ημερήθειας διάταξης. Κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική θάλασσα. Μπόνους. Άννα Ρόσπακ είναι η συγγήτρια. Παρακαλώ παρουσιάστε το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ε, κοιτώ το χρόνο που περνάει. Με την πρώτη ματιά αυτό δεν φαίνεται να είναι προβληματικό θέμα. Δεν είναι, είναι όμως σημαντικό. Το θέμα είναι πρόγραμμα έρευνα, ε, που όπως πολύ σωστά, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Πρόεδρε και ήδη στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς ε, το Κοινοβούλιο στις 29 Οκτωβρίου του 2009 υπέβαλε απόφαση Ε, για ε, νέα μορφή του προγράμματος αυτού σύμφωνα με την συνθήκη της Λισαβόνας. Και τώρα λέγεται το πρόγραμμα αυτό Bonus 169 και αντικαθιστά το Bonus Eranet και Bonus Eranet Plus. Στόχος είναι τα 8 κράτη-μέλη που βρέχονται από τη Βαλτική να συμμετέχουν σε ένα κοινό πρόγραμμα, να ε, επωφελείται το ένα κράτος από τις έρευνες του άλλου και να προωθηθεί η γνώση στον τομέα του περιβάλλοντος ε, και σε άλλους τομείς. Να συγκεντρωθεί η εμπειρογνωμοσύνη. Ε, Δανία, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, Πολωνία, Γερμανία, Σουηδία είναι τα κράτη-μέλη Μέχρι τώρα ούτε τη Λευκορωσία ούτε τη Ρωσία κατάφερα να ε, κινητοποιήσω, να ε, συμμετάσχουν ενεργητικά και οι δύο χώρες αυτές έχουν ποτάμια που χύνονται στη Βαλτική. Δυστυχώς τα ποτάμια αυτά είναι πολύ μολυσμένα και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Γι' αυτό πολύ θα ήθελα να υπάρχει η δυνατότητα συμπερίληψης των δύο χωρών αυτών στο πρόγραμμα αυτό. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Ε, να σας τα πω από μέσα. Συμπεριλαμβάνονται στόχοι, αλλά στόχος είναι να συνδυάσουμε, τις, να συγκεντρώσουμε τις ε, γνώσεις ε, που έχουμε για το τι μπορεί να γίνει με τη βιοπικιλότητα, την ε, αλλαγή του κλίματος, τα ύδατα, τα, οι διαρροές πετρελαίου από πλοία κλπ. Οι πετρελαιοκυλίδες. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντική η γνωμοδότηση αυτή έχω κάποιες τροπολογίες, λίγες, διότι θεωρώ ότι το πρόγραμμα bonus, ότι για το πρόγραμμα bonus δεν θα πρέπει απλά να κινητοποιήσουμε τους ε, συμμετέχοντες, θα πρέπει να τους υποχρεώσουμε να δημοσιεύουν τα αποτέλεσματα των ερευνών τους, ώστε όλοι να μπορούν να επωφεληθούν από την εμπειρογνωμοσύνη, από τις γνώσεις που έχει κάθε χώρα. Αναφέρθηκα στην Λευκορωσία και τη Ρωσία, που είναι τρίτες χώρες. Και τέλος, βρίσκω ότι θα πρέπει εδώ να περιλαμβάνεται και μια επισκόπηση των ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η πρόβλεψη του οικονομικού κόστου τη απώλεια τη ε, βιοπικιλότητα ε, στην ε, Βαλτική. Έχουμε το θέμα του γάδου. Αυτό δεν ισχύει όμω μόνο για το γάδο. Ισχύει και για τον ξηφία, ισχύει και για άλλα ψάρια. Το είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε χρήσιμα αποτελέσματα και πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, ασχοληθούμε από κοινού με το θέμα αυτό. Ελπίζω λοιπόν ότι θα με βοηθήσετε, ε, θα στηρίξετε την ε, μικρή αυτή γνωμοδότηση. Γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν υπήρχαν συναντήσεις με σκιώδεις εισηγητές, αλλά ήταν πάρα πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι αύριο το μεσημέρι. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους λοιπόν να, μου υποβάλουν καλές προτάσεις εδώ και τώρα. Διότι 15-16 Μαρτίου θα πρέπει να κρίνουμε την, έκθεση, την γνωμοδότηση αυτή και θα πρέπει να την στείλουμε για μετάφραση εάν έχουμε ε, περισσότερες τροπολογίες. Πιστεύω ότι είναι θέμα ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Άννα Ρόσπαχ. Πράγματι, η ρήπανση της Βαλτικής είναι θέμα ανησυχητικό. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Να καλωσορίσω μια ε, αποστολή του, από το Κοινοβούλιο της Νορβηγίας. Μιλάμε τώρα για μόλυνση, μόλυνση της Βαλτικής. Ζήτησαν το λόγο αυτοί που μένουν στη Βαλτική, ο Νταν Γιόργενσεν. Ευχαριστώ. Να πω στους ε, καλεσμένους μας από την Νορβηγία ότι βλέπετε υπάρχει ε, χώρο στην αίθουσα. Θα χωρούσαν και νορβηγικά μέλη στην Επιτροπή μας, αν ενδιαφέρεστε. Αλλά καλά, άλλη φορά θα το συζητήσουμε αυτό. να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια, την Αναρόσπαχ. Πιστεύω ότι έχετε βρει πολύ καλή ισορροπία. Φυσικά όταν εμείς εδώ πέρα υποβάλλουμε γνωμοδότηση από την Επιτροπή μας θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην περιβαλλοντική πτυχή και βρίσκω ότι το κάνετε αυτό. Πολύ σωστά. Πρόκειται για τομέα με διασυνοριακά προβλήματα, και εγώ από τη Δανία προέρχομαι όπως και εσείς. Επανειλημμένα χρειάστηκε να εξετάσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών ε, που ε, είναι κάπως επόδυνα για τη Δανία και η Σουηδία και άλλες χώρες ε, νιώθουν τις αρνητικές συνέπειες της ρήπανσης που προέρχεται από τη χώρα μας, ε, για παράδειγμα από, την, ε, από τον τομέα της ε, χειροτροφίας. Είναι ένα από τα προβλήματα της Βαλτικής. Πολύ σωστά μιλάτε για συμπερίληψη και της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, διότι μια σειρά ποταμών γίνονται στη Βαλτική οι χώρες αυτές όμως ε, είναι υπεύθυνε ε, και για μεγάλο μέρος ε, των θαλάσσιων μεταφορών που δημιουργούν προβλήματα. σκοπεύω να υποβάλω κάποιες τροπολογίες, οι οποίες όμως κυρίως αφορούν σύσφυξη κάποιων διατάξεων που εσείς προτείνετε. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε ήδη στην προκαταθική φάση να λαμβάνουμε υπόψη θέματα κλίματος ε, και βιοπικιλότητας. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να γίνεται όσο γίνεται νωρίτερα στη διαδικασία. Και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι κάτι θα πρέπει να γίνεται κατά την ε, φάση της προετοιμασίας. Επίσης δεν ξέρω αν μπορούμε να τονίσουμε διότι στην έκθεση αναφέρονται πολύ λίγα συγκεκριμένα πράγματα για το πώς θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τους διάφορους ε, επιστήμονες και να συγκεντρώσουμε την ε, γνωσιακή βάση που υπάρχει. Είναι πολύ ευγενής ο στόχος, νομίζω συμφωνούμε όλοι, αλλά πολύ λίγο συγκεκριμένο περιεχόμενο υπάρχει εδώ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συμπεριλάβουμε κάτι πιο συγκεκριμένο σε μια γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, αλλά ίσως βρούμε άλλο τρόπο να το κάνουμε αυτό. Πιστεύω επίσης ότι μια και το πρόγραμμα αυτό θα, ε, ε, θα κινείται από πολιτικές ανάγκες, ε, μήπως να μιλάμε και για περιβαλλοντικές ανάγκες ε, και ανάγκες που αφορούν την ε, υγεία. Ε, πάντως γενικά βρίσκω ότι είναι πολύ καλή προσπάθεια και σας ευχαριστώ για τη δουλειά που έχετε κάνει με την εκθεσία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Dan Jorgensen. Ο Dan Jorgensen είπε ότι πράγματι χωράει και η Νορβηγία στην επιτροπή μας, αλλά... καλά, δεν θα ήσασταν τόσο πολύ τότε, αλλά θα ήταν ωραίο αν συμμετείχε και η χώρα σας. Πάντως, καλώς ήρθατε. Τρεις ε, εκθέσεις έχουμε ακόμα. Παρακαλώ λοιπόν προσέξτε λίγο το χρόνο. Δύο λεπτά ε, αναπαρέμβαση. Σα του χάσει. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προτάσεις που κατά την άποψή μου είναι πολύ καλές. Το πρόγραμμα αυτό είναι πάρα πολύ καλό και θετικό. Και ενδεχομένω εδώ στο Κοινοβούλιο θα έπρεπε να τονίσουμε ότι πίσω από αυτό έχουμε την στρατηγική για τη Βαλτική θάλασσα, κάτι το οποίο ήταν μια πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου στην αρχή. Είναι λοιπόν καλό που προχωράει και προοδεύει ακριβώ αυτή η στρατηγική για τη Βαλτική θάλασσα με αυτόν τον τρόπο. Η συγγήτρια ήδη αναφέρθηκε στα περιβαλλοντικά προβλήματα και θα ήθελα να προσθέσω ότι σύμφωνα με τις δικές μου παρατηρήσεις στο Κοινοβούλιο δεν γνωρίζουν όλοι το γεγονό ότι η Βαλτική είναι μια από τις πιο μολυσμένες θάλασσες παγκοσμίω. Θεωρούν πολύ ότι στο βορρά τα πράγματα είναι εντάξει, ότι οι κοινωνίες είναι καλά οργανωμένες, ότι οι πολίτες είναι νομοταγείς και ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σε υψηλό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά όμως η Βαλτική είναι μια από τις πιο μολυσμένες θάλασσες στον κόσμο. Οι προτάσεις της εισηγήτριας νομίζω ότι οι πιο σημαντικές από αυτές αφορούν το γεγονός ότι όλες οι χώρες μέλη της Βαλτικής θα πρέπει να συμμετέχουν στις διάφορες δράσεις και θα ήθελα να διευρύνω κατά κάποιο τρόπο την περίληψη αυτή ώστε να λάβουμε υπόψη μας και τις λεκάνες εκροές στην ε, Βαλτική θάλασσα γιατί μεγάλο τμήμα της μόλυσης προέρχεται από αυτούς τους ποταμούς. Και να πω επίσης ότι σε σχέση με την βιοπικιλότητα και τον υπολογισμό του κόστους θα ήθελα να διευρύνουμε και εδώ πάλι την πρόταση αυτή υπό την έννοια ότι θα πρέπει να να αντιμετωπίζουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τα οικονομικά τους έννοια. Βεβαίως η εξασθένση της βιοπικιλότητας είναι θέμα πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει να το δούμε νομίζω από τη σωστή σκοπιά. Ο κ. Σόνικ. Ευχαριστώ. Αυτό το πρόγραμμα για τη Βαλτική θάλασσα προβλέπει την συμμετοχή και δραστηριότητα οχτών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει και ένα συντονισμό δραστηριοτήτων για την έρευνα για το περιβάλλον και βεβαίω και την ανάγκη αντιμετώπισης κοινών προκλήσεων. Αυτό μας ε, επιτρέπει βεβαίως να διοργανώσουμε τα θέματα έρευνας στην Βαλτική θάλασσα, ξεπερνώντας βεβαίως και φραγμούς οικονομικούς εθνικής φύσης. Κατά άποψή αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική στην Βαλτική θάλασσα, το πρόγραμμα δηλαδή αυτό, και θα ήθελα να πω α, ταχύτατα ποιες είναι οι παρατηρήσεις μου. Έχω κάποιες αμφιβολίες για το μηχανισμό της Κομισιόν σε σχέση με την χρηματοδότηση του προγράμματος στο Real Common Board. Ξεκινάμε την προπόθεση ότι όλες οι χώρες θα καταθέτουν την ε, συνεισφορά τους σε ένα ενιαίο ταμείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για όλα τα προγράμματα. Πώς μπορούμε όμως στη συνέχεια να διασφαλίσουμε ότι η συνεισφορά μιας χώρας μέλους δεν θα καταλήξει σε ένα πρόγραμμα που δεν αφορά την περιοχή του ή τέλο πάντων σε ένα πρόγραμμα δική του αρμοδιότητας υπάρχει κι άλλο ένα θέμα εδώ από την Επιτροπή που λέει ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι χώρες μελή μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια τους για έρευνες, εθνικές έρευνες και τα επιχειρήματα υπέρ αυτού του από αυτής θέσης ποια είναι. Νομίζω ότι στην κάθε χώρα μέλο, δεν επιτρέπουν όλα τα νομικά πλαίσια την ε, καταβολή της εισφοράς σε αυτό το πρόγραμμα. Οπότε γεννάται εδώ το ερώτημα πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το γεγονό ότι τα διάφορα προγράμματα δεν θα επεκταθούν στο δίνικες; Εδώ χρησιμοποιούμε το άρθρο 169 ε, ως βάση. Αλλά έχουμε και άλλα προγράμματα κατά νου όπως αυτά της Eurostat και άλλων, που δεν προέβλεπαν αυτή την ε, χρήση ως μπόνους. Αν προβλέψουμε, αν προβλέψουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία στο πρόγραμμα πλαίσιο, τότε εκ μέρους της Κομισιόν θα έπρεπε να υπάρχει μια λύση που θα διασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος και την ίση συμμετοχή των ενδιαφερόντων. Των ενδιαφερομένων μάλλον, Δεύτερον, η εφαρμογή χρονική του προγράμματος στρατηγική εφαρμογή δύο χρόνια και πενταετής περίοδος μετά από αυτό. Έχουμε όμω κάποιες αφιβολίες, δηλαδή είναι σωστό να υπάρχει μια υποχρέωση για μετάβαση στη στρατηγική φάση. Αυτό νομίζω θα εξαρτηθεί από την πραγματική δυνατότητα που θα έχουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ομολογώ δεν έχω ξαναδεί σε προγράμματα αυτού του είδους. Ευχαριστώ. Μετά τη Δανία, τη Φιλανδία και την Πολωνία, η Λιθουανία ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρόσπαχ για τη θαυμάσια δουλειά που έκανε στην μασία αυτού του εγγράφου. Βεβαίω, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα πρέπει να είναι κοινά και θα πρέπει να υπάρχει κοινή συμμετοχή στην έρευνα για την παρακολούθηση της κατάστασης της Βαλτικής θάλασσας. Είναι καλό να γίνεται αυτό ετησίως και τα πρόσφατα στοιχεία όσον αφορούν την τοξικότητα του περιβάλλοντος δείχνουν ότι η γενική τοξικότητα στη Βαλτική ξεπερνά τα αποδεκτά όρια. Ακόμα και εκεί που σχεδιάζεται να γίνουν μεγάλα έργα υποδομής. Και αυτό μας δείχνει ότι το πρόγραμμα αυτό ο μπόνους, θα πρέπει να αποτελεί μια, μια καθοδήγηση, μια κατευθύντια γραμμή δηλαδή για τους πολιτικούς γιατί θα πρέπει να κάνουμε τα προγράμματα στην ε, Βαλτική και συμφωνώ με την ε, περίληψη, με την συμμετοχή δηλαδή της ε, Λευκορωσίας και άλλων στο πρόγραμμα και σύμφωνα με αυτό που είπε και ο κύριος Σόνικ, θα ήθελα να προσθέσω ότι η σωστή κατανομή των κονδυλίων είναι σημαντική. Οπότε κάποιες χώρες στην Βαλτική λαμβάνουν περισσότερα προγράμματα και νομίζω θα ήταν καλό να διασφαλίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερο δίκη κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των χωρών της Βαλτικής. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για την έκθεση της κυρίας Ρόσπαχ αύριο 25 Φεβρουαρίου και ε, ε, στην Επιτροπή 16 Μαρτίου, εξέταση των τροπολογιών ε, και ε, κατόπιν θα πάει στην, στην Ολομέλεια. Πολύ σύντομα, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που η Βαλτική είναι τόσο μολυσμένη. Ήταν πολύ σωστά τα επιχειρήματα που ακούσαμε, πολύ σωστά μίλησε ο Ντάν για την ε, κτηνοτροφία, την χειροτροφία. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι η Βαλτική είναι κλειστή θάλασσα και αυτό μάλλον είναι το βασικότερο πρόβλημα, διότι ακόμα και αν δεν μολύνουμε τη Βαλτική, το πρόβλημα είναι ότι, για παράδειγμα, αν έχουμε πολύ ε, μακρύ και ζεστό καλοκαίρι, ε, τότε μεγαλώνουν πολύ ε, τα φύκια και κατόπιν αρχίζει και πεθαίνει η θάλασσα. Πάντως, είναι πολύ ευαίσθητη περιοχή η Βαλτική και γι' αυτό θα πρέπει να, φροντίσουμε, να τη φροντίσουμε ιδιαίτερα και γι' αυτό μπορεί μερικές φορές να πληρώσει κανείς για κάποια προγράμματα ε, για τα οποία να μην επωφεληθεί κανείς σε πρώτη, ε, φάση, για παράδειγμα η Πολωνία, ε, αλλά είναι κοινά προγράμματα και η Γερμανία πληρώνει για το πρόγραμμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Φτάνουμε στο σημείο 17 της ημερησίας διάταξης. Ε, κινητοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ε, η συγκίτρια είναι η Τατσιάνα Σάρβου. Της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τεχνολογίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη της ενεργειακής, απόδοσης, που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω δηλαδή ε, μιας καλύτερης κατανομής ενέργειας, βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των μεταφορών. Και τώρα θα σας παρουσιάσω κάποιους από τους σημαντικούς τομείς όπου θα μπορούσαν να βοηθήσουν οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών ώστε να κάνουμε πιο αποτελεσματική τη μετάβαση προς μια ενεργειακή, ενεργειακά αποδοτική οικονομία. Εδώ θα μπορούσαμε λοιπόν να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μην ξεπεράσουν τη ζήτηση. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ευφύ συστήματα ενεργειακά και έναν ευφυή υπολογισμό της ενέργειας ώστε να καταλήξουμε σε εξοικονόμηση. Μετά οι μεταφορές. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών θα μπορούσαν να μειώσουν την ανάγκη για μετακίνηση προσφέροντας ας πούμε τηλεδιασκέψεις, ε, μαθήματα μέσω ίντερνετ και ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να μειώσουμε βεβαίως τις εκπομπές άνθρακα και γενικότερα την μόλυνση ώστε να κάνουμε και, την, ε, και τις μεταφορές πιο ρευστές όσον αφορά και τις μεταφορές των προϊόντων και αγαθών χρησιμοποιώντας πάντοτε τα πιο αποτελεσματικά τα πιο μάλλον αποδοτικά ε, από ενεργειακή σκοπιά οχήματα. Ένα άλλο στοιχείο σχετικό εδώ είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση του κοινού γιατί ένα από τα πιο σημαντικά ενεργειακά στοιχεία εδώ είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά. Πολύ συχνά ο κόσμος κάνει απλά λάθη επειδή δεν είναι ενήμερος. Οπότε αυτό το δυναμικό δεν θα μπορούσε να αξιολογηθεί αν δεν είναι σε θέση οι ίδιοι οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν σωστά αυτές τις τεχνολογίες. Θα πρέπει να έχουμε μια εναρμονισμένη μεθοδολογία για την καταμέτρηση της ενεργειακής απόδοσης επειδή η Κομισιόν επιμένει για το γεγονό ότι για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών θα πρέπει να βρεθεί μια εναμονισμένη τεχνολογία για την καταμέτρηση της ενεργειακής απόδοσης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση να κάνουμε συγκρίσεις βιώσιμες μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ήθελα να σας αναφέρω αυτό το κεφάλαιο που νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό ε, δεν είχα και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου εξάλλου, μόνο μόλις μία εβδομάδα και είχα την έκθεση μόνο στα Ιταλικά. Υπάρχουν και άλλες πτυχές σημαντικές βιβλίες, τις οποίες θα προσθέσω μέσω τροπολογιών και θα καλέσω και τους ε, συναδέλφους να κάνουν το ίδιο. Να λάβουμε όμως υπόψη μας ότι έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πολύ. που ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα, το οποίο έχει σχέση με την προστασία του κλίματος. Κύριε Πνερ. Πρόεδρε, η κυρία Σάρμπου με τρόπο πολύ συνοπτικό μας παρουσίασε τις πτυχές που αφορούν τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών σχετικά με την ανακοίνωση αυτή υπογραμμίζουμε τις ανάγκες και τις δυνατότητε εξέλιξης αυτού του τομέα, βελτιώντας βεβαίως τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και διαχείοντάς τις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Όσον αφορά την τεχνολογική καινοτομία που θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μας στον ενεργειακό τομέα ώστε να μειώσουμε τις εκπομπές, όλα αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ευρώπη να βγει από την κρίση και να καταλήξει σε μια οικονομία πιο ισορροπημένη. Αυτές λοιπόν οι νέες τεχνολογίες μας επιτρέπουν πραγματικά να κάνουμε εξοικονομήσεις ενέργειας σε όλους τους οικονομικούς τομείς και επιτρέπουν επίσης να προσεγγίσουμε αλλαγές και τροποποιήσεις με τον απαραίτητο ρυθμό σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της βιομηχανίας. Μέχρι το 2020 έχει χαράξει φιλόδοξους στόχους η Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε αυτοί οι στόχοι τελικά να υλοποιηθούν και να εφαρμοστούν μέσω μιας κοινή συμφωνίας και να καταλήξουμε τελικά στη μείωση κατά 20% της ε, κατανάλωσης ενέργειας και αντίστοιχα 20% των εκπομπών άνθρακα, όπως επίσης και 20% χρήση ΑΠΕ για την εξοικονόμηση ενέργεια. Η αποτελεσματική λοιπόν χρήση των ενεργειακών πόρων είναι εκ των όνων κάνευ όρος για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Οπότε οι συστάσει που θα πρέπει να δώσουμε θα πρέπει βεβαίω να επικεντρωθούν στον τομέα των κατασκευών, αλλά θα πρέπει γενικότερα να κάνουμε το ίδιο και στον τομέα των μεταφορών, τη στιγμή που αυτό αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό στην γενική κατανάλωση ενέργειας. Οι χώρες μέλη και η Κομισιόν θα πρέπει να ξεκινήσουν μια πρωτοβουλία για αυτό το θέμα. Τώρα, σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, αυτές θα μπορούσαν να αυξήσουν το ρόλο της επιμελητίας στον ε, κλάδο των μεταφορών και θα μπορούσαν πράγματι να μειώσουν τις απώλειες που έχουμε στο εσωτερικό του δικτύου της ε, κατανάλωσης ενεργείας και θα μπορούσαν επίσης να μας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσουμε ευφυεί συστήματα για την ενέργεια στις κατασκευές και αλλού. Όλα αυτά λοιπόν θα έπρεπε να μας οδηγήσουν στο να επηρεάσουμε την συνείδηση των καταναλωτών όταν χρησιμοποιούν αυτή την ε, ενέργεια ώστε να έχουμε τεχνολογίες που θα επιτρέπουν πραγματικά να έχουμε εξοικονομήσει ενέργειας. Και εγώ έχω πρόθεση να καταθέσω τροπολογίε οι οποίε ακριβώ θα τονίζουν το ρόλο των τεχνολογιών και πληροφοριών και επικοινωνιών σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι η μείωση τη χρήση τη ενέργεια και η εξοικονόμησή τη έχει κέριο λόγο στην καταπολέμηση τη μόλυνση του περιβάλλοντο και στην μείωση των εκπομπών, του, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Νομίζω ότι στην ουσία οι τεχνολογίες ε, πληροφοριών και επικοινωνίων έχουν μεγάλο ρόλο στην ε, ενεργειακή απόδοση. Και εξάλλου αυτό αποδεικνύεται από το γεγονό ότι εμείς το θεωρούμε αυτό το θέμα ως προτεραιότητα του εβδόμου ου ε, προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη. Και να καταλήξω λέγοντας ότι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης ιδιαίτερα όσον αφορά τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ιδιαίτερα αναφέρουμε εδώ βεβαίω στην προστασία του περιβάλλοντο και τη υγεία των καταναλωτών όταν χρησιμοποιούμε αυτέ τι τεχνολογίε ακριβώ. Ευχαριστώ. Βιτόριο Πόλη. Πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την παρουσίαση. Σύντομα, θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση που αφορά καταρχήν την εξέλιξη του ηλεκτρικού δικτύου προς ένα δίκτυο FES που θα γνωρίζει δηλαδή και θα είναι σε θέση να συλλέγει την ε, ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βρισκόμαστε ενώπιον της ανάγκης να αυξήσουμε τη συνολική απόδοση της χρήσης της ενέργειας και να μεγιστοποιήσουμε την συμβολή των ΑΠΕ. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς να χρησιμοποιήσουμε σε μεγάλο βαθμό και με τρόπο πεπισμένο και πιστικό τις ε, τεχνολογίες αυτές πληροφοριών και επικοινωνιών. Από την άποψη αυτή λοιπόν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε εις βάθος και τα συστήματα συμπαραγωγής που διανέμονται ώστε να αυξήσουμε με τον τρόπο αυτό τη συνολική απόδοση του ενεργειακού συστήματος. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό επειδή ακριβώς μέσω της συμπαραγωγής διανομής ενέργειας που θα λειτουργεί ταυτόχρονα με τη χρήση φυσικού αερίου και φυσικού αερίου και ε, βιοαερίου θα μπορούσαμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα αποθήκευσης του αερίου ώστε να έχουμε μια ευελιξία στο δίκτυο του αερίου και σε τελική ανάλυση να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία και στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο μέσω μιας πιο γενικευμένης χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Και τέλος θα ήθελα να υπογραμμίσω μεταξύ των πολλών πτυχών που αναφέρθηκαν το ότι θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε την ατομική κινητικότητα με μια εικονική κινητικότητα. Αυτό που θα μπορούσε ας πούμε να συμβεί και εδώ στο κοινοβούλιο μας. Δηλαδή να έχουμε λιγότερες συνεδριάσεις, ενδεχομένως ε, μεγαλύτερες διάρκειας, αλλά με την εξαποστάσεως χρήση των τεχνολογιών για την προετοιμασία των ε, συζητήσεων μέσω τηλεδιασκέψεων που τώρα πια είναι μια πραγματικότητα παντού. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά όχι πάντα. Είναι ωραίο να έχει κανείς μπροστά του το πρόσωπο και να μην έχει μόνο μέσω οθόνη μια τηλεδιάσκεψη. Ωραία στο Ρώση. Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι για το 17, 18, 19 δεν έχουμε το κείμενο στα Ιταλικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι απαράδεκτο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απαράδεκτο να μην έχει τα κείμενα αυτά στην Ιταλική γλώσσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η προθεσμία για τις τροπολογίες στην περίπτωση 17 είναι αύριο και στο 19 οι, τροπολογίες, η προθεσμία είναι αύριο, 18 1 Μαρτίου πολύ κοντά, για το 16 είχαμε το κείμενο στα τελικά, αλλά και, και πάλι η προθεσμία για τις τροπολογίες ήταν αύριο. Πρόεδρε, σας καλώ λοιπόν και να προσθέσω και κάτι άλλο για τα βιοκτώνα, σημαντικό θέμα που συζητήσαμε προηγουμένως. Άκουσα από εσά και την συγγήτρια ότι επεκτείνοντας και παρατείνοντας τους χρόνους για την κατάθεση των τροπολογιών, διατρέχουμε τον κίνδυνο να μην έχουμε στη διάθεσή μας όλες τις τροπολογίες. Εμείς εδώ δεν παίζουμε, είμαστε στο Κοινοβούλιο. Σας καλώ λοιπόν θερμά μέσω του Προεδρείου, μέσω του Προέδρου του Κοινοβουλίου, αφού λείπουν οι διερμηνές, να τους προσλάβετε. Εμείς τις θέλουμε τις μεταφράσεις, αφού έχουμε κάθε δικαίωμα να τις έχουμε. Να προσέχετε λοιπόν και να αναλάβετε τα απαραίτητα μέτρα. Αν λείπουν μεταφραστές, να τους προσλάβετε. Ναι, μέχρι μεθαύριο θα την παρατείνουμε, αλλά περισσότερο δεν γίνεται, διότι πρόκειται για νομοδότηση προς την Επιτροπή Βιομηχανίας και θα ψηφίσει. Ε, και είτε θα το κάνουμε γέρος ή θα πάει στο καλά στον αχρήστον η πρότασή μας. Δυστυχώς λοιπόν ε, δεσμευόμαστε από την επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή. Η επιτροπή μας όμως πρέπει να ομορφωνομοδοτήσει διότι μας αφορά το θέμα. Σας παρακαλώ λοιπόν για την κατανόησή σας. Ε, και έχουμε τόσες γλώσσες εργασίας, η Νορβηγία δεν συμμετέχει ακόμα στην Ένωση, τότε θα είχαμε άλλη μία, αλλά θα είχαμε τότε 23 γλώσσες που θα έπρεπε να μεταφραστούν. Μπάρμπαρα Τεμπρίν, θέλετε το λόγο? Όχι. Α, παρεξήγηση ήτανε. Το Τσάνα Σάβο. Δεν θέλει το λόγο. Να κλείσουμε λοιπόν τη συζήτηση αυτή. Προθεσμία 25 Φεβρουαρίου για τις τροπολογίες ε, το μεσημέρι. Το επόμενο θέμα είναι το θέμα του Κοσλοτούι. Χρηματοδοτική συνδρομή της κοινότητας για τον παροπλισμό των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού Κοσλοτούι στη Βουλγαρία. Η Αντώνια Παρβάνοβα έχει αναλάβει την έκθεσή μας. Ε, της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια έκθεση σχετικά με την πρόταση για ένα κανονισμό του Συμβουλίου για να επιτεθεί η οικονομική βοήθεια όσον αφορά τις μονάδες 1-4 ε, του σταθμού του Κοσλοντούι. Και θα έπρεπε να σας πω εδώ ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Δεν υπήρχε χρόνος για να προετοιμαστεί η γνωμοδότησή μας, η οποία συμφωνεί με την, ε, σύμφωνη με την Επιτροπή ΙΤΡΕ Και ζητώ συγγνώμη που δεν είχα χρόνο να ε, να φροντίσουν να μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Γι' αυτό ε, η έκθεση έχει συνταχθεί στα αγγλικά και προσβλέπω στην ανταλλαγή απόψε με τους σκιώδεις συζητητές και θα έπρεπε να πω ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε όλες ε, τις, ε, όλους τους σκιώδες που πρότειναν οι ομάδες. Αυτή η έκθεση λοιπόν θα πρέπει να υποστηριχθεί από την Επιτροπή MD με βάση δύο συλλογισμούς. Πρώτα απ' όλα η πολιτική αλληλεγγύης και ίσης μεταχείρισης μεταξύ κρατών μελών, όπως το πρόγραμμα τη Λιθιονίκης Σλοβακία, όπως και η υποστήριξη για τη Βουλγαρία που τελειώνει το 2009 και δεύτερον το 2006 αποφάσισε η κυβέρνησή μας να περάσει σε άλλη στρατηγική και να διαλύσει τη μονάδα άμεσα με βάση οικονομικούς παράγοντες και παράγοντες ασφαλείας ώστε η χώρα να μπορεί να διαπραγματευτεί ε, ε, μια νέα συμφωνία ή συμμεταχείριση μέχρι το 2014 ε, για να εξασφαλίσει μια διάλυση ασφαλή. Η Επιτροπή υποστηρίζει επιπλέον οικονομική υποστήριξη για δεκατομμύρια ευρώ μεταξύ δύο δραστηριοτήτων, 60% των χρημάτων για ε, την των δραστηριοτήτων, 40% για, για μέτρα ε, αντιμετώπισης των ενεργειακών μέτρων, για να αντισταθμίσει την απώλεια ε, ικανότητας παραγωγής. η επέκταση της βοήθειας κοινότητας είναι απαραίτητη για να πραγματοποιηθούν οι στόχοι κυρίως για να εξασφαλιστεί η ασφαλής διάλυση της μονάδος, εξασφαλίζοντας προστασία περιβάλλοντος και διαφάνεια. Και υπογραμμίζω το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της συμμετοχής του κοινού. Η, η γνωμοδότηση βασίζεται στους κανόνες ασφάλειας και περιβάλλοντος σύμφωνα με τον κανονισμό για την προστασία των εργαζομένων και του κοινού κατά της ακτινοβολίας και πρόσβαση στις πληροφορίες, συμμετοχή του κοινού και διαφάνεια για να ληφθούν οι, οι αποφάσεις που είναι κατανοητές. Επέκταση οικονομικής βοήθειας για μέτρα που χρειάζονται στον ενεργειακό τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, στις τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές και στην τροφοδοσία ε, του κοινού κυρίω ε, όσον αφορά το κλείσιμο των σταθμών 1 έως 4. Υπογραμμίζεται η οικονομική βοήθεια, αλλά και η συνοχή με τη στρατηγική ενέργεια και περιβάλλοντο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητεί περιεκτική προσέγγιση και λήψη υπόψη των συνεπειών από το κλείσιμο των τεσσάρων πυρηνικών σταθμών. Οι τέσσερις σταθμοί οδήγησαν στην εφαρμογή των κυρίων αρχών, επί των οποίων η κοινοτική στρατηγική βασίζεται και νομίζω ότι πρέπει η Επιτροπή μας να την υπογραμμίσει. Πρόκειται για την ε, μείωση των εκπομπών ε, αερίων θερμοκηπίου, ε, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, την ασφάλεια τροφοδοστησίας και η ικανότητα παραγωγής θα πρέπει να αντισταθμιστεί με εισαγωγές πρωτογενούς ενέργειας και με ενέργεια ορυκτή εσωτερική, θα ήθελα να σας προσθέσω ορισμένα στοιχεία. Θεωρείται ότι η απώλεια ικανότητας ενέργειας λόγω της ε, πρόορης ε, παύση λειτουργίας αυτών των αντιδραστήρων θα οδηγήσει σε, σε περιορισμό της έκκληση αριών του θερμοκηπίου για την περίοδο 2011-2013 και θα έχουμε περίπου 1,2 γίγκα ε, γραμμάρια γίγκα και θα έχουμε 18.000 κιλοτόνους ε, οξυδίου του άνθρακα που θα εξοικονομηθούν. Και ε, ο οι επιπτώσεις για τα γειτονικά κράτη είναι πολύ σημαντικές. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθηθεί η μείωση του διοξιδίου του άνθρακο και οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Τέλο, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η οικονομική διαχείριση του προγράμματο μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι σύμφωνη με του οικονομικού ε, κανονισμού και του εφαρμοστικού κανόνε και ευθύνη μα είναι ω Δημοσιονομική Αρχή να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια ε, και θα προβλεφθούν στον ε, προπολογισμό του προσεχούς έτους και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι διαδικασίες ε, που θα εφαρμοστούν. Υπογραμμίζοντας η Επιτροπή δεν έχει τηρήσει τους κανόνες, κυρίως το άρθρο 53 Δέλτα και το άρθρο 43 6, το οποίο έχω περιλάβει στην έκθεσή μου για την περίοδο 2010-2013. Βεβαίως θα πρέπει πρώτα ε, ε, ε, να ακολουθήσουμε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικοδόμησης, αλλά θα πρέπει η Επιτροπή να λάβει τα μέτρα ώστε να περιληφθεί αυτός ο κανονισμός. Τέλος, η θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει πλήρη εφαρμογή των ενεργειακών στρατηγικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η οικονομική βοήθεια να οδηγήσει ε, στην άριστη εφαρμογή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Παρβάνοβα. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό στη Βουλγαρία, αλλά είναι σημαντικό και για του γειτόνου σα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εδώ η συγγήτρια της Επιτροπής Ήτρε, η Ρεμπέκα Χάρμς. Παίρνει τον λόγο λοιπόν για τους πρασίνους ή εκ μέρους της Ήτρε. Παρακαλώ. Συχνά οι πράσινοι έχουν καλές ιδέες και γι' αυτό αποφάσισαν όχι μόνο να είμαι εισηγήτρια στην Επιτροπή Βιομηχανίας, ε, αλλά να συνεργαστώ, ε, να ασχοληθώ εδώ πέρα με την ε, σκιώδη εισήγηση στην Επιτροπή σας. Έτσι, αυτό απλοποιεί τα πράγματα, γίνονται, μπορεί να αποφύγει κανείς τις αντιφάσεις και να φτάσουμε πιο εύκολα σε ένα κοινό παρονομαστή. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι πρέπει διαπιστένουμε ότι ο παροπλισμός ε, του Κοσλοντούι ε, για τα τμήματα 1 έως 4 είναι σωστή απόφαση. Οι τεχνικοί λόγοι που παρουσιάστηκαν ε, ήταν ότι είναι ακόμα χρήσιμη, δεν υπάρχει δυνατότητα επισκευής ο πρόωρος παροπλισμός ε, θα ε, συμβάλλει όχι μόνο, στην ασφάλεια όχι μόνο στην ε, Βουλγαρία αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες χώρες. Όπως το βλέπω εγώ, οι μονάδες 1, 2, 3, 4 Ε, παροπλίζονται πέντε χρόνια προτού να έπρεπε να γίνει αυτό ούτως ή άλλως για τεχνικούς λόγους. Μιλάμε λοιπόν για μια πενταετία, μπορεί να μιλάμε και για έξι ή εφτά. Πιστεύω ότι με αυτή τη βάση το συνολικό ποσό που ε, μετεβάζεται στην ε, Βουλγαρία και που προέρχεται από τον ε, που προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 860 εκατομμύρια μέχρι το 2013. Αυτό αποτελεί πολύ καλή συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνέπεια της σύστασης για παροπλισμό των μονάδων. Για μένα παραμένει το θέμα τι θα γίνει με τα χρήματα που θα δοθούν ε, στην τελευταία δόση. 300 εκατομμύρια ευρώ προβλέπεται να διατεθούν και το ποσό αυτό θα πρέπει να μοιραστεί σε δύο διαφορετικά ποσά. 180 εκατομμύρια θα δοθούν για περαιτέρω άμεσες εργασίες που θα πρέπει να γίνουν ε, πριν τον παροπλισμό των μονάδων 3 έως 4 και για την ε, ασφαλή ε, αποθήκευση των αποβλήτων κλπ. Αυτό δεν είναι λίγο διότι οι προϋποθέσεις μέχρι τώρα στη Βουλγαρία για προσωρινή αποθήκευση δεν μπορεί να περιγραφούν ως καλές. Έτσι, λίγο προσεκτικά λέω στους συναδέλφους ότι θα μπορούσατε να το βελτιώσετε αυτό και ε, εμένα μου έκανε εντύπωση ως ιδιαίτερο πρόβλημα ότι για την ε, τελική αποθήκευση δεν έχουν ε, ληφθεί καθόλου μέτρα και τα στοιχεία καύσης ε, που ε, προκύπτουν από το Κοσλοτούι ε, εξάγονται προς τη Ρωσία. Αυτό δεν αποτελεί συμβολή στην καλύτερη ασφάλεια ούτε στην Βουλγαρία ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο μάλλον στη Ρωσία. Είναι προβληματικός τρόπος διάθεσης των αποβλήτων αυτών και δεν συμβάλλει στην αποτελεσματική λύση ε, του θέματος των πυρηνικών. Και άλλωστε η ανακύκλωση δεν έχει καμία σχέση με την τελική αποθήκευση. Ε, θέλω να πω στην εισηγήτρια και το έχω πει και σε βουλγάρους συνάδελφους, ε, τα 300 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να δοθούν στη Βουλγαρία, να χρησιμοποιηθούν για νέες κατασκευές. Τα 120 εκατομμύρια όμως που είχαν προβλεφθεί για την δημιουργία εναλλακτικών πηγών ενέργειας που δεν ορίζονται σαφέστερα όμως. Αυτά τα 120 εκατομμύρια θα πρέπει να ε, αποταμιευθούν σε ένα ταμείο ώστε η Βουλγαρία να λάβει μέτρα σχετικά με, την, ε, με τον παραπλησμό και την τελική αποθήκευση των ε, αποβλήτων. Έχω ασχοληθεί με το θέμα αν η Βουλγαρία επιγόντως χρειάζεται βοήθεια για την δημιουργία εναλλακτικών ε, δομών παραγωγής ενέργειας. Κατά τη γνώμη μου, η ε, ε, αυτάρκεια της, Ρουμανί... της Βουλγαρίας δεν αποτελεί καθόλου πρόβλημα. Η Κομισιόν στην πρότασή της αναφέρει ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου το σύνολο της περιφέρειας. Δεν υπάρχουν σημαντικές, δεν υπάρχουν πολλές γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. και δεν μπορεί στόχος ε, των ε, πληρωμών αυτών ενισχύσεων ε, για το Κοσλοντούι, δεν μπορεί στόχος των πληρωμών αυτών λοιπόν να είναι να προωθήσουμε δομές παραγωγής να είναι οι δομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία που θα εξάγεται σε μη ορισμένες γειτονικέ χώρες. Ε, πόσο μάλλον όταν οι δομές όταν οι δομές που παίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας χρησιμοποιούν είτε λιγνίτη είτε έχουμε την άλλη την ε, ε, ατομική ε, μονάδα παραγωγής ενέργειας. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Διακόπτη. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέτε, αλλά είναι πολλά θέματα τα οποία θα κρίνει η Επιτροπή ε, Βιομηχανίας. Ευχαριστώ πολύ. Η Κάριν Κάντενπαχ, ε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του ε, συναδέρφου μου που δεν μπορεί να παρευρεθεί και γι' αυτό θα ήθελα ε, το πρώτο μέρος της παρέμβασής μου ε, να το αφιερώσω στις δικές του θέσεις. we είναι σωστή απόφαση της, του παραπλησμού αυτών των μονάδων. να Λαμβάνοντα υπόψη ε, ότι θα χρησιμοποιηθούν και οι ανθρώπινοι πόροι ε, για την διαδικασία παροπλισμού και αυτό θα έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις και κοινωνικές. Θα καταθέσουμε τι τροπολογίε μα ε, και θα υπογραμμίσουμε τις περιβαλλοντικές πτυχές. Επίσης, υποστηρίζουμε την πρόταση της κ. Παρανόβα για τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα και την παρακολούθηση των πόρων μα. Αυτή είναι η θέση του σκιώδου συγητή μας. Ε, θα ήθελα όμως ε, και ως ε, Αυστριακή να πω προσωπικά ότι χαίρομαι όταν παροπλίζονται ατομικές μονάδες και και ότι βρίσκω θλιβερή την απόφαση της Βουλγαρίας να συνεχίσει να επενδύει στην πυρηνική ενέργεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ισαπίνε Βίλς. Είμαι σκιώδη εισηγήτρια για την ΚΟΕ για την έκθεση αυτή να συμφωνήσω με την παρέμβαση της συναδέλφου Χάρμς. Συμφωνούμε με την ε, χρηματοδότηση για παροπλισμό των μονάδων 3 ε, και 4, ε, για θέματα διάθεσης των, της διάθεσης των αποβλήτων. Ε, αυτά δεν θα πρέπει να επανεξάγονται σε χώρες ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας. Το θέμα είναι οι εναλλακτικέ δομέ παραγωγή ενέργεια. Θα θέλαμε όμω οι σχετικοί πόροι να διατεθούν για ε, προγράμματα ανανεώσιμης ενέργειας, ε, αύξηση της αποτελεσματικότητας ε, της ενέργειας και της ασφάλειας τροφοδότησης. Θα ήθελα επίσης να κάνω την εξής παρατήρηση. Η ασφαλής διάθεση ατομικών αποβλήτων δεν υπάρχει, ωστόσο θα πρέπει να διαθέσουμε σωστά τα υπάρχοντα απόβλητα και βρίσκω σημαντικό να τονίσουμε ότι η Βουλγαρία συνεχίζει να εξάγει ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης σημαντικό είναι αυτό που είπε η κυρία Χάρμς και που αναφέρεται στην έκθεση της Ήτρε. Ο παροπλισμός των μονάδων 3 και 4 είναι οριστικός και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να ξαναλειτουργήσουν οι μονάδες αυτές. Είναι σημαντικός λοιπόν ο παροπλισμός των μονάδων αυτών. Όσον αφορά την διαφάνεια κατά τη διάθεση των, ε, ε, των χρηματικών πόρων τα 300 εκατομμύρια δηλαδή αυτά πώς θα ε, διατεθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο παρελθόν έχει επενδύσει σε ε, λογικά προγράμματα, σε καλά προγράμματα ε, παραγωγής ενέργειας στην Βουλγαρία. Τα χρήματα αυτά τελικά όμως έχουν διατεθεί για μονάδες που χρησιμοποιούν λιγνίτη, για παράδειγμα ή σε ατομικές ε, εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να εξεταστούν τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από την Κομισιόν η κυρία Πλαουμχίπερ. Να μας παρουσιάσετε τις θέσεις σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που στηρίζει την πρότασή μας Βρίσκουμε πολύ καλό το ότι στηρίζεται και τους δύο πυλώνες και τον ατομικό όσον αφορά την ε, διάθεση των αποβλήτων και τον ε, τομέα της ενέργειας. Ε, θα ήθελα να πω το εξής. Από το Ταμείο Παροπλισμού δεν έχουμε στηρίξει ούτε μονάδες λιγνίτη, ούτε μονάδες ατομικές, ε, αποκλειστικά ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ε, προγράμματα αποτελεσματικότητας της ενέργειας, ε, διότι ακριβώς αυτά τα προγράμματα παρουσιάζουν πολύ γρήγορα αποτελέσματα σε σχέση με άλλα μεγάλα προγράμματα. Γι' αυτό πιστεύουμε από πλευρά της Κομισιόν ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό το παράθυρο αυτό προς τη Βουλγαρία τουλάχιστον μέχρι το 2012 και να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε προγράμματα αποτελεσματικότητας ενέργειας καθώς και σε δίκτυα διότι αν αφαιρέσουμε τέσσερις, πυρηνικούς, ε, τέσσερις πυρηνικές μονάδες από τα δίκτυα θα αλλάξει η ισορροπία ε, στη Βουλγαρία και θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις ε, διότι τα μέσα που είχε η Βουλγαρία δεν αρκούσαν για κάτι τέτοιο έχουμε ε, επενδύσει μαζικά σε προγράμματα διάθεσης ε, των ε, αποβλήτων διάθεσης απορριμμάτων και δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα για τις ενεργειακές επενδύσεις. Θα παρακαλούσα να ακολουθήσετε την πρότασή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βλαμφίπερ. Η συγγήτρια για να κλείσει παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω βουλγαρικά. Ευχαριστώ πολύ για όλες ε, τις συνεισφορές σας. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που κάνετε και τα σχόλια. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την υποστήριξή της σχετικά με τη διαφάνεια και για τα θέματα που έχουν σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα. και για τα κεφάλαια το οποία θα διαθέσει η Βουλγαρία. Μερικέ διευκρινήσει πριν από τον παροπλισμό των μονάδων η Βουλγαρία εξήγαγε ηλεκτρικό ρεύμα ε, της των 2.000 γιγκαβάτ. Μετά από τον παροπλισμό των μονάδων Νιώθηκαν οι εξαγωγέ στι γύρω χώρε, δηλαδή Γαλλία, Μακεδονία, Αλβανία, ε, με Ελλάδα, ε, Μακεδονία, Σερβία. Για αυτό το λόγο η χώρα μας τώρα δεν συζητάει την επαναλειτουργία των μονάδων, αλλά μιλήσαμε για το 2009, για τις μονάδες 2 και 3, να αντιμετωπιστεί η μεγάλη κρίση, η μεγάλη εξάρτηση ή όταν υπάρχει πρόβλημα με τροφοδοσία σε αέριο, ε, τα προβλήματα Ρωσίας και Ουκρανίας. Αλλά δεν έκανε μια τέτοια πρόταση η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν υπάρξει μια τέτοια κρίση στο μέλλον, η επαναλειτουργία δεν είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται. Συνεπώς, η Βουλγαρία δεν ισχυρίζεται ότι ποτέ θα λειτουργήσουν πάλι αυτές οι μονάδες. Τώρα, η διευκρίνηση την οποία θα ήθελα να κάνω είναι η εξή. Η Βουλγαρία έχει μία σύμβαση με τη Ρωσία για τα καύσιμα. Τώρα, όσον αφορά το καύσιμο από τις μονάδες 1, 2, 3, αυτή η σύμβαση είναι ακόμα ενεργή. Αλλά θα χρησιμοποιηθούν για λιγότερο ε, επικίνδυνα απόβλητα που θα προέρχονται από την εγκατάσταση ε, που αφορά τα κτίρια. Συνεπώς η Βουλγαρία δεν εξαρτάται και δεν θα εξα... Ε, από αυτό το καύσιμο και δεν θα εξαγάγει αυτό το καύσιμο. Λοιπόν, τα χρήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό τα απόβλητα, τα οικοδομικά απόβλητα αν θέλετε, θα αποθηκευθούν σε αυτούς τους χώρους με ασφάλεια. Ακόμα ένα σχόλιο. Έχει σχέση με, αυτά τα 2.000 γιγκαβάτ και την αντικατάστασή τους. θα καλυφθούν από προϊόντα άνθρακα. Θα πρέπει να κλείσουμε τέσσερις εγκαταστάσεις ε, που λειτουργούν με κόκ. Εάν κλείσουν θα έχουμε blackout στη χώρα μας, θα έχουμε προβλήματα ή θα έχουμε ηλεκτροδότηση διακεκομένη, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρξει αποσταθεροποίηση της ε, τροφοδότησης ενέργεια, της ηλεκτροδότησης δηλαδή στη χώρα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντικατασταθούν αυτά τα 2.000 γιγκαβάτ, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα και να μην ε, καταφύγουμε σε τεχνολογίες που είναι επιβλαβείς ε, για το περιβάλλον. Με τα χαράς θα ήθελα να συζητήσω με το σκιώδη συγγητή τα θέματα αυτά, ώστε να καταλήξουμε σε μία συνένεση την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία είναι 1η Μαρτίου. Λοιπόν, στο τέλος της εβδομάδας θα μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. 1η Μαρτίου. Το μεσημέρι είναι η καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Και η νέα διαδικασία κατάθεσης τροπολογιών ισχύει και για αυτή την έκθεση. Ας περάσουμε τώρα στο τελευταίο θέμα της σημερινής μας συνεδρίασης, της πρωινής συνεδρίασης, η εξουσία εκχώρησης νομοθετικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έγινε μια αλλαγή. Το Κοινοβούλιο έχει περισσότερες αρμοδιότητες ε, όσον αφορά ε, τις αρμοδιότητες ε, προς την Επιτροπή. Η διάσκεψη των Πρόεδρων πρότεινε ότι ως Κοινοβούλιο να εγκρίνουμε την έκθεση στην Ολομέλεια. Η Νομική Επιτροπή είναι υπεύθυνη επί της ουσίας και συχνά τα θέματα αφορούν την Επιτροπή μας. Γι' αυτό θα πρέπει να ετοιμάσουμε μια γνωμοδότηση. Παρουσίασα αυτή τη γνωμοδότηση στα αγγλικά μόνο. Θέλουμε να είμαστε σε ίσης όρις με το Συμβούλιο Υπουργών και όχι όπως ε, στην επιτροπολογία του παρελθόντος να βρισκόμαστε σε μια νυχτική θέση. Επίσης, να έχουμε αρκετό χρόνο για να μπορούμε να αξιολογήσουμε την ε, αντιπροσωπεία. Στις ε, θερινές διακοπές, στις χρονιάτικες διακοπές, οι καταστάσεις είναι διαφορετικές. Όπως και το Συμβούλιο και εμείς θέλουμε να συμμετέχουμε στις εργασίες της Κομισιόν. Ε, δεν μπορούμε να λέμε στους ε, εθνικούς επιρογνώμονες ότι επήγει το θέμα και τελικά το Κοινοβούλιο να μην ε, συμμετέχει καιρό στις εργασίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν διοργανική συμφωνία ανάμεσα στην, ε, στο Συμβούλιο, το, την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο, διότι είναι θέματα τα οποία αφορούν και τα τρία θεσμικά όργανα. Αυτά πολύ σύντομα για τη σύσταση της Επιτροπής μας. Ο Πέτερ Λίζε ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όχι μόνο που μου δίνετε το λόγο, αλλά και για τη δουλειά σας. Ο πρόεδρος μας ήταν στην προηγούμενη θητεία, ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Θεμάτων. Ε, θεώρησα λοιπόν ότι ήταν καλό να αναλάβει τη δουλειά αυτή, διότι είναι θέμα που έχει να κάνει με την επιρροή του Κοινοβουλίου και την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας προς όφελο των πολιτών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρότασή σας αυτή. Γενικά περιέχει τα βασικά σημεία. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί διότι πολλές ε, από αυτές τις ε, πράξεις δευτερεύουσας ε, νομοθεσίας, δευτερογενούς νομοθεσίας, δευτερογενούς δικαίου, μπορεί να προσπερνούν την Επιτροπή μας. Έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό στα πλαίσια της έκθεσης της Μπάρμπαρα Ντεμπρύν. Γενικά, Μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις προτάσεις του Προέδρου. Ε, κάποιες μικρές διευκρινήσεις στο σημείο 1. Θα θέλαμε να προσθέσουμε από πλευράς του ΕΛΚ ότι το δευτερογενός αυτοδίκαιο ε, θα πρέπει να εξετάζεται ανάλογα με το θέμα που αφορά, διότι συχνά οι πράξεις αυτές μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Στο σημείο 4 προτείνω να μην μιλάμε για early approval, αλλά για urgent procedure, για επίγουσα διαδικασία, αντί για έγκαιρη έγκριση. Γενικά, χρειαζόμαστε χρόνο να εξετάσουμε τα θέματα αυτά. Όταν Επειδή το θέμα θα πρέπει να μπορεί κανείς να ξεφύγει από τις προθεσμίες που έχουν οριστεί. Στο σημείο 5, στην τελευταία παύλα, λέμε να καλεί το Κοινοβούλιο σε προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις ε, που ε, οργανώνονται σε σχέση με αυτά τα delegated acts, τη, τη δευτερογενή νομοθεσία. Να πούμε involving parliament που συμπεριλαμβάνει το Κοινοβούλιο στη, στην προκατακτική εργασία, στην προπαρασκευαστική εργασία, διότι δεν γίνονται μόνο συνεδριάσεις, ανταλλάσσονται και ηλεκτρονικά μηνύματα. Ε, αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα το οποίο τόνισε και ο Πρόεδρος πρέπει να έχουμε σαν στόχο το Κοινοβούλιο να μην έχει χειρότερη θέση από το Συμβούλιο και αυτό ισχύει για το σύνολο της διαδικασίας αυτής. Πρόκειται για μικρές ε, προτάσεις βελτίωσης. Ε, γενικά βρίσκω πολύ καλή την ε, πρόταση του Προέδρου μας και θα συμφωνήσουμε με αυτήν. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι δεν υπάρχουν πολύ ισχυρές γνώμες στο θέμα αυτό. Οι συντονιστές περισσότερο έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Πέτερ Λίζε. Το urgent procedure, η επίγουσα διαδικασία, είναι άλλη διαδικασία από την έγκαιρη ε, ε, ε, έγκριση. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην προκαλέσουμε σύγχυση αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Το involving in preparatory work είναι σίγουρα καλύτερα από το να καλεί το Κοινοβούλιο να συμμετέχει στις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις. Αυτό το βρίσκω πολύ καλό. Και στο σημείο 1, εμείς είπαμε in principle, καταρχάς, η παλιά διαδικασία επιτροπολογία θα αντικατασταθεί από τη νέα διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 290. Μήπως προσθέσουμε εδώ κατά περίπτωση να γίνεται σχετική εξέταση. Προθεσμοί για την ε, υποβολή τροπολογιών είναι μεθαύριο 25 Φεβρουαρίου στις 12. Φτάσαμε στο τέλος της ε, ημερήσιας διάταξης για το πρωί. Θα συνεχίσουμε στις 3 με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε στη ημερήσια διάταξη. Λήξη της συνεδρίασης. Κάνει τη δουλειά. So.